Good morning, ladies and gentlemen. I reopen the meeting of the Budgetary Control. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου του προϋπολογισμού. Πρώτο θέμα είναι η Γεωργία. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο, τους Γενικούς Διευθυντές, τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ξεκινώντας να δώσω το λόγο τον ε, κύριο Νίσαλα από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Παρακαλώ. Ε, Mr. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, αγαπητέ Επίτροπε, είναι με μεγάλη χαρά για μένα να παρουσιάσω την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2010 για το θέμα των δαπανών ως προς τη γεωργία το περιβάλλον, τις θαλάσσιες επιθέσεις, την αλία, την υγεία και την προστασία του καταναλωτή. 56,8 δις ευρώ είναι το ποσό που αντιστοιχεί σε όλα αυτά τα θέματα, 45% των πληρωμών του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2010. Στην παρουσίασή μου θα επικεντρωθώ στη γεωργία και στην ανάπτυξη της υπαίθρου. πολιτικές που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων για τη Γεωργία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανάπτυξη της Υπέθρου. Το πρώτο ταμείο υπάγεται στον πρώτο πυλώνα. Τα βασικά μέτρα είναι το σύστημα ενιαίας πληρωμής και άλλα ε, προγράμματα άμεσων ενισχύσεων δαπάνες για την ανάπτυξη της υπαίθρου εντάσσονται στο δεύτερο πυλώνα. Και, το, ο δεύτερος πυλώτα, πυλώνας ε, καλύπτει πληρωμές για λιγότερο ευνοημένες περιοχές, για επενδύσεις σε ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για υποδομές σε, σε αγροτικές περιοχές. Αυτά που βρήκαμε, τα ευρήματα για το 2010, θέτουν τέσσερα θέματα. Πρώτον, ε, η συμμόρφωση με το τυπικό των διαδικασιών από πλευράς συναλλαγών. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την, τον άμεσο έλεγχο των συναλλαγών. Διενεργήσαμε λοιπόν άμεσες δοκιμές ελέγχους σε 208 συναλλαγές. 87 από αυτές παρουσίαζαν ένα ή περισσότερο σφάλμα. Ο τελικός αντίκτυπος του ποσοτικοποιημένου σφάλματος εκτιμάται στο 2,3%. Πάνω δηλαδή από το κατόφλι ε, της ουσιαστικότητας. Η έλεγχοι του ελεγκτικού συνεδρίου επιβεβαίωσαν τη συχνότητα των σφαλμάτων. Και μάλιστα επιβεβαίωσαν ότι αυτή η συχνότητα δεν κατανέμεται με ισότιμο τρόπο. Ως προς τον πρώτο πυλώνα, είχαμε να κάνουμε κυρίως με σφάλματα ακρίβειας. Ε, κυρίως ε, δηλώσεις μεγαλύτερων εκτάσεων από αυτές που υπήρχαν στην πραγματικότητα. Και είχαμε και σφάλματα επιλεξιμότητας. Επίσης, κάποιες παρατηρήσεις για τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου. Μιλούμε ε, για το σύστημα ΕΑΝΤΑΣ, Άγιαξ όπως γνωρίζετε. Είδαμε ότι έχουμε μία ακριβή στοιχεία στις βάσεις δεδομένων και ατελείς διασταυρώσεις. Ας πάρουμε μία συγκεκριμένη βάση δεδομένων, το σύστημα εντοπισμού και ταυτοποίησης των αγροτεμαχίων. Η χρήση είναι απαξιωμένη θα έλεγα. Όλες αυτές οι βάσεις δεδομένων περιλαμβάνουν εκτάσεις που δεν είναι επιλέξιμες, όπως για παράδειγμα βραχώδεις εκτάσεις ή δάση. Σε γενικές γραμμές είχαμε και πληροφορίες που ήταν απαξιωμένες τελείως. Όλα αυτά έχουν ε, αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα των διασταυρώσεων. Μιλούμε λοιπόν για τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου. Για τα οκτώ αυτά συστήματα, βάσει του Άγιαξ, πρέπει να γίνουν έλεγχοι επιτόπου τουλάχιστον στο 5% των δικαιούχων. Είδαμε λοιπόν ότι οι έλεγχοι αυτοί δεν διενεργούνται σωστά βρήκαμε εσφαλμένες μετρήσεις και καθυστερήσεις στους ελέγχους από πλευράς των ε, ελεγκτικών αρχών των κρατών μελών. Είδαμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα κόστη που ζητούνταν δεν συνοδεύονταν από το κατάλληλο υλικό τεκμηρίωσης. Και η τέταρτη παρατήρηση έχει να κάνει με το την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης για τη Γεωργία το 2010. Το 2009 η έκθεση είχε επιφυλάξεις για, τα, για τις δαπάνες που είχαν να κάνουν με τον άξονα 2 για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Το 2010 η Επιτροπή αποφάσισε να άρει τις επιφυλάξεις αυτές. Με βάση την ανάλυση που έχουμε κάνει, η απόφαση αυτή δεν είναι καθόλου δικαιολογημένη. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με βάση όλα αυτά, το ελεγκτικό συνέδριο συμπεραίνει ότι, ότι τα ουσιαστικά ασφάλματα είναι σημαντικά. Ό,τι έχει να κάνει με το σύστημα Άγιαξ δεν περιλαμβάνει ουσιαστικά σφάλματα. Εκεί μιλούμε για 40 ε, δις ευρώ οι δαπάνες για την ανάπτυξη της υπαίθρου είναι εκτεθειμένες σε μεγάλο βαθμό σε σφάλματα. Υπάρχει δηλαδή εκεί μεγάλος ε, ε κίνδυνος. Παρά πολλά, τα πολλά χρόνια των ουσιαστικών βελτιώσεων στα συστήματα παραμένουν ουσιαστικοί κίνδυνοι ως προς την, ε, το τυπικό και τη συμμόρφωση με το διατακτικό όλων αυτών των πληρωμών. Και όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στη δουλειά μας. Βασικό είναι να βελτιώσουμε το σύστημα Ajax, να περιλαμβάνει δηλαδή στοιχεία ενημερωμένα και αξιόπιστα. Τέλος, ποιες είναι οι συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου. Θα πρέπει λοιπόν η Επιτροπή να αναλάβει δράση ώστε το σύστημα εντοπισμού και ταυτοποίησης των αγροτεμαχίων να ενημερώνεται τακτικά. Προτείνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι αρχές πληρωμών θα ε, κάνουν τη δουλειά τους και θα συμπληρώσουν τα κενά ε, που αφήνει το σύστημα εντοπισμού αγροτεμαχίων. Τέλο, η ποιότητα των ελέγχων επιτόπου από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βελτιωθεί ούτως ώστε να εντοπιστούν αξιόπιστα οι περιοχές οι οποίες δεν είναι επιλέξιμες. Κύριε Πρόεδρε, ο συνεισηγητής, ο ήταν υπεύθυνο για το δεύτερο πυλώνα. Είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσει πληροφορίες. Και εγώ είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω ε, σε οποιαδήποτε ε, ερώτηση τυχόν ε, τεθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ο Επίτροπος Τσιόλος παρακαλώ. Θα θέλατε να απαντήσετε στις παρατηρήσεις του δικαστηρίου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, αξιότιμοι εκπρόσωποι του ελεκτικού συνεδρίου. Η σωστή διαχείριση των ε, κονδυλίων βάσει της κοινή γεωργικής πολιτικής είναι βασικός στόχος για μένα. Προσπαθήσαμε να, το, ε, να κάνουμε το παν. Μιλούμε για τις προόδους που έχουν σημειωθεί φέτος. Πιστεύουμε ότι 2,3% είναι το συνολικό ποσοστό σφάλματος. Για το ΦΕΟΓΑ το ποσοστό αυτό είναι κάτω του 2% και για τις άμεσες πληρωμές είναι ακόμα μικρότερο αυτό το ποσοστό. Σίγουρα το ελεκτικό συνέδριο παρουσιάζει ένα πιο ε, ψηλό ποσοστό κινδύνου, ωστόσο και αυτό βαίνει μειούμενο. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι γίνεται σε γενικές γραμμές σωστή διαχείριση αυτής της ε, πολιτικής έχουμε ενισχύσει το ρόλο των οργάνων πιστοποίησης, ώστε οι διαβεβαιώσει των κρατών μελών να είναι ακόμα πιο στεναρέ και να μην υπόκεινται σε αμφισβητήσεις, κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στις ανησυχίε του ελεκτικού συνεδρίου. Έχουμε ε, βασιζόμαστε σε στατιστικές ελέγχους, σε στατιστικά στοιχεία ελέγχου που μας δίνουν τα κράτη-μέλη και καλούμε τις αρχές πιστοποίησης να κάνουν δειγματοληψία. Τρία κράτη-μέλη έχουν δοκιμάσει αυτό το σύστημα φέτος και άλλα δύο κρατημέλη θα το κάνουν του χρόνου. Κάναμε και διάφορες άλλες δράσεις για να βελτιώσουμε ε, την ποιότητα των ε, συστημάτων ελέγχου ως προς το Άγιαξ. Έχουμε για τις άμεσες πληρωμές ε, ποσοστό σφάλματος της τάξης του 1%, του 1%. Τα, οι χώρες με τα περισσότερα προβλήματα ήταν η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Πορτογαλία février Στην ετήσια έκθεση βλέπουμε ε, ότι ε, όντως μπαίνουν με τα, τα ποσοστά αυτά. Έχουμε μια αποστολή ελέγχου το 2011 στη Ρουμανία ως προς τη Βουλγαρία λοιπόν το σχέδιο δράσης ε, οριστικοποιήθηκε στα τέλη του Νοεμβρίου του 2011 και αυτό έχει επιβεβαιωθεί από μια αποστολή ελέγχου πριν από δύο εβδομάδε. Κατά τη διάρκεια του 2012 θα έχουμε και άλλε αποστολέ ελέγχου και για τη Ρουμανία και για τι άλλε χώρε. Η Γενική Διεύθυνση για την ε, Γεωργία έχει καταθέσει επιφύλαξη για την ε, Πορτογαλία και ζήτησε την εφαρμογή ενό ενισχυμένου σχεδίου δράση. Θεωρεί λοιπόν η Επιτροπή ότι στι αρχέ του 2012 θα οριστικοποιηθεί αυτό το σχέδιο δράση Αν δεν έχουν ολοκληρωθεί εργασίε μέχρι το τέλο αυτή τη ε, προθεσμία και μάλιστα με τη σωστή ποιότητα, θα ζητήσω να ε, υιοθετηθούν όλες οι απαραίτητες διατάξεις για να προστατευτούν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, ε, θα ε, υιοθετηθούν όλες οι όλα τα απαραίτητα μέτρα για τις χρηματοδοτικές διορθώσεις. Προκειμένου όμως να έχουμε σωστή πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες του συστήματος, θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να κάνουν μια σε βάθος ετήσια αξιολόγηση ως προς την βάση δεδομένων για την ε, γεωργία. Αυτό το οποίο είπε δηλαδή το μέλος του ελεκτικού συνεδρίου. Εάν σημειωθούν και εμφανιστούν αδυναμίες, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν διορθωτική δράση. Το 2010 ήταν μια πιλωτική χρονιά και θα έχουμε πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα λίαν συντόμως. Τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε τη σωστή διαχείριση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω τέσσερα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης που προτείναμε εμείς ως Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η μεταρρύθμιση αυτή θα συμβάλλει στη βελτίωση του συστήματος και θα μειώσει ακόμα περισσότερο το ποσοστό του σφάλματος. Μιλώ για την ενίσχυση του ρόλου των αρχών πιστοποίησης, οι οποίες ε, παίρνουν σωστή δειγματοληψία, κάνουν τη σωστή δειγματοληψία όλων αυτών των συναλλαγών. Προτείνουμε να γίνει αυτό υποχρεωτικό για όλα τα κράτη-μέλη από το 2014 και μετά. Με διτό στόχο, πρώτον, να έχουμε ε, σιγουριά για την ποιότητα των ελέγχων των κρατών μελών και από την άλλη μεριά, βέβαια, να εστιάσουμε του ελέγχου εκεί που είναι περισσότερο απαραίτητοι. Και στη συνέχεια μπορούμε να μειώσουμε ε, του ελέγχου εκεί όπου το ποσοστό σφάλματο είναι αποδεκτό έτσι ώστε να δοθεί και κίνητρο στα κράτη-μέλη να μεριμνήσουν περισσότερο για τους ελέγχους αυτά τα ίδια και θα ενισχύσουμε ε, το σύστημα των πληρωμών ούτω ώστε να υπάρχουν, ε, να γίνονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι ανακτήσεις. Αντί για το τωρινό 50% προτείνουμε να δίδεται το 100% ε, των ποσών που δεν έχουν ανακτηθεί και θα έχουμε αναστολή πληρωμών σε περίπτωση αμέλειας. Τρίτον, προτείνουμε την απλούστευση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Σημερίζομαι ε, τη σημασία που δίδετε εσείς και το ελεγκτικό συνέδριο. Για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις προτείνουμε να υπάρχει μια ε, πιο ελαφριά διαδικασία, να ενοποιηθούν και να απλωστευθούν οι κανόνες της αιρεσιμότητας. Για τις πληρωμές που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της υπαίθρου, θέλουμε να βασιστούμε ε, σε σύστημα καταποκοπήν, εφάπαξ, βάση στάνταρ κόστους. Τέταρτη πρόταση της μεταρρύθμισης είναι η έννοια του ενεργού, του δραστήριου αγρότη στη μεταρρύθμιση θέλουμε να έχουμε άμεσες ενισχύσεις μόνο στους ενεργούς αγρότες, να εξαιρεθούν δηλαδή οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ασκούν γεωργική δραστηριότητα οι ίδιοι ή που την ασκούν μόνο στο περιθώριο άλλων δραστηριοτήτων τους. Η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, ε, είναι αντικείμενο της συναπόφασης. Έτσι η δική σας Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού ε, θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ελπίζω και βασίζομαι στη βοήθειά σας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και παραμένω στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ερώτημα. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ο πρώτος που θα κάνει σχόλια και θα θέσει ερωτήματα είναι ο εισηγητής ο κύριος Φέλνερ. Mr. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την δική, μας τη δική μου ευγνωμοσύνη <laughs> στο Ελεκτικό Συνέδριο και στην Επιτροπή. Διότι σήμερα νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας ε, μία ε, βάση για μία πολύ καλή συζήτηση τα θέματα αυτά που αφορούν τα πάνε που γίνεται το τομέα που μας αφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να θίξω τέσσερα θέματα. Πρώτα απ' όλα, ανάπτυξη πέθρων, το παράδειγμα το οποίο μας, τις εξαιρέσεις τις οποίες δίνει το ελεκτικό συνέδριο για τις ε, λιγότερο επιτροπές και πρασίνισμα της ΚΑΠ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να κάνω ένα γενικό σχόλιο το οποίο απευθύνεται στο ε, ε, ελεγκτικό συνέδριο. Διαβάζοντας το 355 λέει ότι οι πληρωμές έγιναν με κάποιες ε, αριθμητικά σφάλματα. Αυτά είναι κακά νέα. Απ' την άλλη, αργότερα βλέπω το ελεγκτικό συνέδριο ότι παρόλα αυτά άμεσες πληρωμές που κάλυξαν την δεν είχαν αριθμητικά λάθη. Καλό νέο είναι αυτό. Όταν τα διάβασα όλα αυτά, κάπως μπλέχτηκα, διότι δεν κατάλαβα τα πράγματα. Οι άμεσες πληρωμές είναι της τάξης του 43 δις, το 77% δηλαδή των δαπανών. Και ακόμη, και κοιτώντα έτσι, έχουμε την εντύπωση ότι το 77% φαίνεται να αποτελεί εξαίρεση από τον κανόνα κατά κάποιο τρόπο. Μ' αρέσει να είναι το bulldog, αυτός που επαγρυπνεί, που εποπτεύει το ελεκτικό συνέδριο. Αλλά έχω την εντύπωση, και αυτό δεν μου αρέσει, ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι θα έπρεπε να. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, είναι επιτυχές το σήμερα. Είμαστε σε θέση το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων να δούμε ότι πραγματικά δεν εμπεριέχεται του αριθμητικά λάθη. Αλλά νομίζω ότι το 77% είναι τέτοιο ποσοστό που δεν θεωρείται εξαίρεση του κανόνα. Το, το αντίθετο. Θα μπορούσε να κάνει ένα σχόλιο από αυτό το ελεκτικό συνέδριο. Τώρα, η πρώτη παρατήρηση. Η ανάπτυξη ήθελες παρά το γεγονός λοιπόν ότι κάποια θέματα γίνονται ε, με σωστό τρόπο, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι 12 δις θεωρείτε ότι δεν έχουν γίνει σωστά. Λέει στην απάντησή της Επιτροπής στην παράγραφο 356 ότι θεωρεί ότι το εποπτικό σύστημα βελτιώνεται συνέχεια και θα ε, επιληθούν τα προβλήματα και μειώνει το ποσοστό του σφάλματος σε αυτό το τομέα. Βεβαίως, το προφανές το είναι ποιο είναι το ποσοστό σφάλματος την περιοχή, ώστε να κατανοήσουμε περί τίνος πρόκειται. Δεν ξέρω αν ο Επίτροπο Τσόλο θα μπορούσε να μα δώσει μια απάντηση. Θα ήταν ενδιαφέρον όμω να δούμε πραγματικά ποιο είναι το ποσοστό σφάλματο στον τομέα αυτό. Και βεβαίω, το Ελεκτικό Συνέδριο συμφωνεί με το γεγονό ότι έχουμε δει πολλέ φορέ ότι υπάρχει βελτίωση συνεχής και λογικά θα αναμέναμε στον τομέα αυτό μείωση του ποσοστού σφάλματος. Και Προσπαθούμε να ζούμε σε έναν κόσμο χωρίς λάθη. Εάν λοιπόν βελτιώνεται η κατάσταση συνεχώς όπως λέει η Επιτροπή, κάποια στιγμή θα πρέπει να υλοποιήσουμε το στόχο μας. Πότε πιστεύει η Επιτροπή ότι δεν θα χρειάζεται πλέον να ανησυχούμε για τέτοιου σφάλματα. Ποια είναι τα μέτρα το αναφέρατε ακροθυγώς κύριε Επίτροπε, αλλά για την επόμενο ε, δημοσιονομικό πολιετές πλαίσιο, τι μέτρα πιο συγκεκριμένα προτείνετε, μπορείτε να πτύξετε το θέμα. Κάτι άλλο που αφορά επίσης την ανάπτυξη πέθρου. Χθε συζητήσαμε εκτενώς με τον Επίτροπο Χάν το θέμα των ε, διαφροντικών μείων και κατά κάποιο τρόπο αυτό εν μέρη εξηγεί γιατί το ήταν εκτεθειμένο σε τέτοιο μεγάλο κίνδυνο το Περιφερειακό Ταμείο. Δεν έχω ακριβείς αριθμούς ποσοστών σφαλμάτων, ούτε για την ανάπτυξη της υπαίθρου, ούτε για το Περιφερειακό Ταμείο. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη, πολύ μεγάλη διαφορά εδώ. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον να μας πει η Επιτροπή πώς συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί, διότι είναι πιο αντικειμενικέ μετρήσει που αφορούν την ανάπτυξη τη υπαίθρου και θα πρέπει, ε, ε υποκειμενικά, με συγχωρείτε, αντικειμενικά, συγγνώμη, και θα πρέπει να τα μετρήσουμε. Είναι θέμα κυρώσεων, όπως λέγεται χθε. Μπορεί η Επιτροπή κατά κάποιο τρόπο να επιβάλλει κυρώσεις στα κράτη-μέλη. Ή το νομικό πλαίσιο, ή διαφορετική φιλοσοφία διαχείριση των θεμάτων αυτό από τις διάφορες γενικές διευθύνσεις οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα και τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να συνάγουμε συμπεράσματα και να μάθουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ήπιαμε καφεδάκι με τον κύριο Πέτρο προηγουμένω και συζητήσαμε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το θέμα των κυρώσεων. Α μα πούνε όλοι λοιπόν και άλλοι. Στον τομέα αυτό τη ανάπτυξη του Πέθρου, πώ λειτουργεί το σύστημα τη επιβολή κυρώσεων. Διότι πιστεύω ότι είναι σημαντικό οι κυρώσει να είναι κάτι το οποίο να αισθάνονται ότι επιβάλλονται τα κράτη. Τώρα, ανέφερε τα σχήματα, το ελεγκτικό συνέδριο, τα σχήματα ενίσχυσης και προγράμματα ενίσχυσης προβλέπονται για τα περισσότερα. Και επέκρινε το όλο σύστημα εδώ και πολύ καιρό ακόμη και στην ειδική έκθεση του 2009 το ελεκτικό ότι το σχήμα αυτό, το πρόγραμμα αυτό δεν εξασφαλίζει την πλήρη διαφάνεια και την σωστή αναλογία κόστους κόστους-οφέλους. Πιστεύετε ότι τέτοιου είδους και αυτή είναι η ερώτησή μου στον Επίτροπο Τσόρος. Πιστεύετε ότι το θέμα αυτό μόνο και μόνο σε αυτή την περίπτωση μόνον και η μεταφορά του βουτύρου που ανέρχεται σε τόσα εκατομμύρια είναι ανισχυτική. Δηλαδή συμμερίζεται από αυτό που λέει το ελεκτικό συνέδριο ότι δεν υπάρχει πάντα σωστή αναλογία κόστους κόστους-οφέλους. Μπορείτε να μας πείτε για ποιο τρόπο πιστεύετε ότι θα πρέπει αυτό το θέμα, το ειδικό να το προσέξουμε ιδιαίτερος. Και γιατί σας προκαλεί τέτοιο πονοκέφαλο. Επίσης, στην απάντηση της Επιτροπής διάβασα ότι η Επιτροπή πεπισμένη ότι αυτό ήταν ένα επίσημο σφάλμα το οποίο διαπιστώθηκε εδώ και υπάρχουν και άλλοι τομεί στους οποίους βλέπω ότι τέτοιου είδους σημαντικά θέματα δεν συζητούν ούτε Ελληνικό συνέδριο, ούτε η Επιτροπή με το κράτη-μέλη τα ενεχόμενα. Τριμερός. Επίτροπος Τσόλος. Επίτροπε Τσόλος και ε, ελεγκτικό συνέδριο. Πιστεύετε ότι μία τέτοια τριμερή συνεδρίαση θα μπορούσε τέτοιου είδους ε, διστάμενες απόψεις να τις έχουμε αποφύγει και να μην συμβαίνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν. payments have to be recovered from by the member states authorities. As regards the system of recoveries at member state level, the court recently concluded a special report. Τώρα, σε μία ειδική έκθεση της ε, ελεκτικού συνεδρίου βλέπουμε ότι όλη η διαδικασία έχει βελτιωθεί, αλλά θα πρέπει κάποιοι κανόνες να αποσαφινιστούν περαιτέρω, ώστε να μην δίδονται διαφορετικές ερμηνείες και δημιουργούν, και μεταξύ. Έχω την εντύπωση ότι προβλέπετε κάποιες αλλαγές στα πλαίσια της πρότασης ε, της πράσινης ΚΑΠ 2020. Έχετε την εντύπωση τελικά ότι τα κράτη-μέλη ανακτούν ε, τα ποσά τα οποία έχουν ε, δοθεί στους δικαιούχους που δεν τα δικαιούνταν τελικά. Σε ποιο επίπεδο μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κύριε Επίτροπε, μπορείτε επίσης να μας πείτε ποια είναι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί σε αυτή την πρόταση που έγινε για να βελτιωθεί το σύστημα. Και προς το ελεκτικό συνέδριο πιστεύετε ότι τα μέτρα αυτά είναι επαρκή. Θα είναι επαρκή. Δεν μίλησα τώρα για το πρασίνισμα της ΚΑΠ. Άκουσα ότι η ΚΑΠ θα πρασινίσει στο μέλλον. Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και χαίρομαι. Απ' την άλλη όμως, δυσκολεύουν τα πράγματα. Γίνεται πιο πολύπλοκο το σύστημα και η αυξανόμενη ε, πολυπλοκότητα του όλου συστήματος ίσως δημιουργήσει και κινδύνους ε, μεγαλύτερους. Δεν πιστεύετε ότι οι μηχανισμοί θα είναι πολύ πιο πολύπλοκοι και όσον αφορά την ε, σωστό τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται οι ρυθμίσεις θα είναι τα πράγματα δύσκολα. Κύριε, κύριος Χατζημαρκάκης, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα σε σχέση με την παρουσία των συναδέλφων. Να πω ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν τόσο πολύ λίγοι συνάδελφοι παρόντε τη στιγμή την οποία κάνουμε τον έλεγχο του πιο σημαντικού μέσου του προβλησμού. Η ομάδα μου χαίρομαι διότι εκπροσωπείται σωστά. Αλλά ειλικρινά δεν είμαστε πολλοί, αλλά όλοι εδώ είμαστε. Θα ήθελα το θέμα αυτό λοιπόν να το τονίσω, δεδομένου ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό σε σχέση με τους φορολογουμένους που εκπροσωπούμε. Θα ήθελα όπως πέρσι κύριε Τσόλες, να σας δώσω εύσημα, διότι υπάρχει πραγματικά βελτίωση συνεχιζόμενη. Πολύ καλό είναι αυτό, διότι έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε πώς έχουν τα πράγματα επακριβώς. Υπάρχουν ε, παρόλα αυτά κάποια προβλήματα για την ε, ανάπτυξη της Πέτρου και είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε κάποια πράγματα σωστά, όπως και στα θέματα συνοχής και της περιφερειακής ανάπτυξης. Αλλά υπάρχουν θετικά σημεία για βελτίωση. Όσον αφορά τώρα τις ερωτήσεις που θέλω να σας κάνω, θα ήθελα να μιλήσω για την ανάκτηση. Και εδώ πρέπει να πω ότι σωστά βλέπω να γίνονται τα πράγματα, χαιρετίζω τη διαφάνεια και βρίσκω ότι τον... είχατε και πολύ καλές ανακοινώσεις προς τον τύπο Καλυσίας. Είπε τον Οκτώβριο ότι και για τα χρήματα τα οποία ζητήσατε να ανακτήσετε 40 εκατομμύρια, ποιε χώρε αφορώνται εδώ. Αυτού του είδου η διαφάνεια μα βοηθά να βρούμε πού είναι τα προβλήματα και βοηθά και τα κράτη-μέλη την επόμενη φορά να μην εγγραφούν σε αυτόν τον μαύρο πίνακα, σε αυτόν τον κατάλογο. Βοηθά να βελτιωθούν τα πράγματα και σα ευχαριστώ γι' αυτό. Όμω πάλι με την ανάκτηση υπάρχουν προβλήματα. Και σε αυτά τα προβλήματα έχουμε ιδιαίτερη διασύνδεση με το ότι η ανάκτηση σε διαφορετικά χρονικά σημεία συμβαίνει στα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει ενιαίος κατάλογος ρυθμίσεων πότε θα γίνει μια τέτοια ανάκτηση. Υπάρχει και ο κανόνας των 50%. Όμως τα αριθμητικά στοιχεία από τα κράτη-μέλη δεν είναι πάντα συγκρίσιμα. Το ελεγκτικό συνέδριο σε μια ειδική έκθεσή του μας έδωσε θετική βάση εργασίας. Οι τόκοι με μη ενιαίο τρόπο εισπράττονται η χρονική στιγμή της ε, καταχώρησης ε, του αιτήματο είναι πάντα διαφορετική και αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις οικονομικά και φυσικά επιπτώσεις αρνητικές για μας, για την κοινότητα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει καθυστερημένη κίνηση της ε, ε, υλοποίηση της ανάκτησης από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό για τα κράτη-μέλη χρειαζόμαστε σαφέστερους κανόνες, ακόμα πιο σαφείς κανόνες, με σαφείς προθεσμίες. Να τεθεί προθεσμία μέχρι πότε τέτοιου είδους ε, αχρεωστήτως καταβληθέντα θα μπορούν να ανακτώνται και πρέπει να έχουν ανακτηθεί. Χρειαζόμαστε ρυθμίσεις για τους τόκους που απουσιάζουν. Σας ερωτώ πότε θα υποβάλλετε τις ενιαίες ρυθμίσεις για τους τόκους και τις ρυθμίσεις για τις ανακτήσεις ένα άλλο θέμα αφορά τις παλαιές, ε, τα παλαιά ε, ζητήματα ανάκτησης από την αρχή της ε, δεκαετίας του 2000. Είναι μεγάλα αυτά τα ποσά, δεν ήταν τόσο αποτελεσματικές οι διαδικασίες ανάκτησης όπως σήμερα. Τίθεται το ερώτημα, τι θα κάνουμε με αυτές τις παλαιές απαιτήσει Κύριε Πίτροπε, πριν από εσά είχε δημιουργηθεί μια task force για την ανάκτηση. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίε εντωμεταξύ. Υπάρχει αξιολόγηση καθοριστική τι θα πρέπει να γίνει και τι πρέπει να συμβαίνει με αυτέ ε, τι ανακτήσει. Ίσως μια επικοδομητική λύση να βρούμε για τι παλαιέ αυτέ απαιτήσει. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Chairman. Um... Σε ευχαριστώ πρόεδρε. Και πάλι για άλλη μια φορά θέλω να τονίσω ότι συζητούμε αυτά τα πράγματα εδώ χωρίς να έχουμε κάποιο παρόντα από το Συμβούλιο, καθότι γνωρίζω. Παρότι φυσικά είναι τα κράτη-μέλη από πλευρά του που κάνουν τις περισσότερες δαπάνες αυτών των μεγάλων ποσών κονδυλίων που διατίθενται. Συνεχίζω να τονίζω αυτό το διαφθορτικό πρόβλημα που εξακολουθούμε να έχουμε στις διαδικασίες απαλλαγής, χωρίς απαλλαγή. Κάποιες παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω σχετικά και αφορούν κυρίως τον ρόλο των κρατών μελών. Και γι' αυτό επικεντρώνομαι με τέτοιο τρόπο και ένταση όσον αφορά το Συμβούλιο σε αυτό το θέμα. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά την διακρύβωση ατυπιών όσον αφορά τα κράτη-μέλη τα ίδια, την ανείχνευση τέτοιων παρατυπιών. Αν αληθεύει από ό,τι γνωρίζω, είναι ευθύνη των κρατών μελών να ανοιχνεύουν τέτοιου είδους παρατυπίες αν δούμε όμως τον πίνακα εδώ, στην σελίδα 76, στη σημείωση 6 παράτημα 1, και δούμε όσον αφορά το τι γίνεται σε σχέση με την πιστοποίηση ε, για τις ε, παρατυπίες βλέπουμε τεράστιες διαφορές μεταξύ αυτών που δηλώθηκαν από τα κράτη-μέλη και αυτών που ζητήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στο τέλος-τέλος. Διαρωτώ με πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένα τέτοιο μεγάλο χάσμα, μεγάλο κενό μεταξύ αυτών που ανοιχνεύουν τα κράτη-μέλη για τα ίδια τα κράτη-μέλη που αφορώνται και αυτών που διακριβώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος τέλος ότι ίσχυε. Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ 14 εκατομμυρίων και 460 εκατομμυρίων. Μπορεί να υπάρχει μια μικρή διαφορά, έστω να το δεχτώ, αλλά τέτοιες τεράστιες διαφορές τελικά δεν είναι εύκολο να γίνουν κατανοητές. Εκτός αν ένα κράτος μέλος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του για αυτή την ανείχνευση. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι διαδραματίζουν σωστό ρόλο από πλευρά σου στα κράτη-μέλη για την ανείχνευση τέτοιων ε, παρατυπιών. Άλλο ερώτημα, το επόμενο. Ο τρόπος με τον οποίο <clears throat> τα κράτη-μέλη ε, χρηματοδοτούν τα ε, χρήματα τα οποία θα έπρεπε να ανακτηθούν. 90% από τα ίδια τα κράτη-μέλη, από δημόσια κονδύλια γίνεται αυτό. Αντί να υπάρχει ανάκτηση από τους τελικούς ε, αποδέκτες και ε, όσους ωφελήθηκαν τελικά. Και αυτό είναι πάλι κάτι το οποίο δεν κατανοώ. Γιατί πώς να το αποκαλέσω, δεν είναι κάτι το παράνομο, αλλά είναι αξιοπερίεργος τρόπος να αντλούνται, ε, να δίνονται επιπλέον κονδύλια στον γεωργικό τομέα, πέρα από τα τεράστια κονδύλια τα οποία δαπανούμε είδος, ήδη από κρατική πλευρά σε αυτόν τον τομέα για τη γεωργία, δεν μπορούμε να ανακτήσουμε από τους ε, εποφεληθέντες ε, ε, δικαιούχους τελικά. Δηλαδή ο φορολογούμενος, οι πολίτες πληρώνουν για την ανάκτηση από πλευρά ενό κράτους. Να το κάνουμε με γενικό κανόνα, να πούμε ότι είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο. Χρήματα τα οποία καταβάλλονται σε ένα γεωργό αχρεωστήτο θα πρέπει από αυτό να επιστρέφουν μέσω ανάκτησης και όχι μέσω του εθνικού κορβανά του κράτους μέλους. Και η τελική μου ερώτηση αφορά το περιβάλλον όσον αφορά τα προγράμματα για τη γεωργία. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την γραπτή της απάντηση. Όμως πρέπει παρόλα αυτά να πω ότι ακόμα περισσότερο περιπλέκεται η υπόθεση προσπαθώντας να βρούμε την άκρη. Στην γραπτή μου ερώτηση επικεντρωνόμουν στην ε, ειδική έκτακτη έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για τα προγράμματα αγροπεριβαλλοντικά, όπου λέει το ελεγκτικό συνέδριο ότι είναι τόσο περίπλοκα και τόσο δύσκολο να αξιολογηθούν, να αποτιμηθούν, που δεν είναι δυνατό να μετρήσουμε αν επιτυγχάνουμε τους στόχους που θέλουμε να επιτευχθούν ή όχι. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με αυτό το πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω, να σας ρωτήσω πέρα από όλα όσα μας υποβάλατε στα στοιχεία της γραπτής σας απάντησης, να σας ζητήσω να αποσαφηνίσετε τι γίνεται σε σχέση με αυτό. Ζητώ συγγνώμη, πρέπει να πάω να ψηφίσω στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 10. Ίσως θα πρέπει λοιπόν να απουσιάσω πρωτού απαντήσει ο Επίτροπος. Σε σχέση με την ε, παρουσία εκπροσώπων των κρατών μελών που δεν είναι διαθέσιμη, Όμως η γραμματεία του Συμβουλίου πλήρως ε, σημειώνει αυτά τα οποία αναφέρονται. Έτσι λοιπόν τα κράτη-μέλη θα πληροφορηθούν κατά λεπτός για αυτά τα οποία ε, διαβουλευόμαστε εδώ. Αυτά σε σχέση με αυτό και το τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα ο κύριος Στάς θα λάβει τον λόγο. Η ομάδα του είναι λοιπόν έτσι πλήρη. Ehm, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα στην ερώτησή μου, στην παρέμβασή μου, τρία θέματα να καλύψω. Καταρχήν, τα προβλήματα όσον αφορά την δημοσιοποίηση του ε, πίνακα του καταλόγου των τελικώς επωφεληθόντων. Συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Έχει δώσει μεγάλη μάχη η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή ώστε να υπάρχει συνολικός κατάλογος των επωφελούμενων όσον αφορά τα διαθετικά ταμεία, το Ταμείο για τη Γεωργία ένας τέτοιος ε, πίνακας, ένας τέτοιος κατάλογος θα έπρεπε να είναι διαθέσιμος όσο αφορά τους πολίτες μας, να δημοσιοποιείται. Όμως υπήρξε μια απόφαση του 10 του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λόγω λέει προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι αυτή τη στιγμή ανέφικτο, αδύνατο να δημοσιοποιηθεί ο κατάλογο ο πίνακα των τελικώς επωφεληθέντων. Ερώτησή μου, ποια διαβήματα και βήματα θα κάνετε εσεί στο Συλλογικό Σώμα των Επιτρόπων ω επίτροπο, ώστε να ανταποκριθείτε σε αυτή την απόφαση τη νομολογία του 10 αλλά να δοθεί ε, ή δυνατόν συνέχεια στο αίτημα και να υπάρξει δημοσιοποίηση κατασκευή καταλόγου αυτών των υποφεληθέντων. Δεύτερο, αφορά και τον ίδιο τον Επίτροπο για την Γεωργία το ερώτημα αυτό. Εισαγωγικά είπε όμω ε, το μέλος ε, του ελεγκτικού συνεδρίου και ευχαριστούμε γι' αυτό ποιε προσπάθειες αναπτύσσονται ώστε ο έλεγχος ο έλεγχος όλων αυτών των ε, δράσεων να μπορεί να παρακολουθείτε και αναφέρθηκε έλεγχη επιτόπου, δορυφορικά συστήματα, Πολύ καλά όλα αυτά. Είναι τμήμα του, της διαδικασίας θεματολογικά της χορήγησης απαλλαγής. Από την άλλη όμως πλευρά έχουμε και κενά, ελλείψεις. Καλή δημοσιονομική έλεγχη είναι η μία πτυχή έλεγχοι όσο αφορά παρατυπίες. Αλλά έχουμε, πρέπει να έχουμε και ελέγχους για την αποτελεσματικότητα της χρήσης των κονδυλίων για τη γεωργία. υπάρχει τέτοια εποπτεία, τέτοιος έλεγχος για την βέλτιστη χρήση και το αποτέλεσμα, την αποτελεσματικότητα αυτών των δράσεων. Και σε μια εκπομπή της φλαμανδικής τηλεόρασης τηλεοπτικών συνεργείων πήγαν στην Πράγα με συγχωρείτε, πήγαν στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μίλησαν με πολλούς γεωργούς και διαπίστωσαν στη Θράκη ότι υπήρχε ένα πρόβλημα όσον αφορά τις ε, επιχορηγήσεις ε, μεταξύ παλαιών και νέων γεωργών. Αναφέρεται ότι μέσω του συστήματος ε, επιδότησης και εδώ λόγω της καλλιέργειας βάμβακα έχουμε αρνητικές επιπτώσεις γιατί δεν υπάρχει πραγματική πρόσβαση σε αυτές τις επιχορηγήσεις. Γιατί, διότι οι παλαιοί γεωργοί, οι πιο ηλικιωμένοι γεωργοί έχουν την κυριότητα αυτών των εκτάσεων και αν θέλετε είναι μια ρύθμιση για το δικό τους εισόδημα. Ε, έτσι γίνεται αδύνατο για τους νέους γεωργούς που καλλιεργούν αυτά ε, τα τα φυτά να έχουν πρόσβαση στις επιχορηγήσεις. Βλέπουμε αυτή η ηλικιωμένη γεωργή είναι, ένα, είναι πάνω από 55. Αυτό είναι όμως πρόβλημα και νέοι θα πρέπει να μπορούν να ασχοληθούν με τη γεωργία στην επαγγελματική τους αυτή σταδιοδρομία. Μια τελευταία ερώτηση. Η ποιότητα των επιχορηγήσεων, των ενισχύσεων. Τι κάνετε εσείς για να βελτιωθεί κάπως η υπόθεση. Είχα αναφέρει, αναφέρθηκε τώρα το βαμβάκι. Αλλά ερώτηση Προ προς το ελεγκτικό συνέδριο. Έχετε επαρκείς ελέγχους, ελέγχετε επαρκώς την υπόθεση. Για τους ελέγχους που έγιναν το 2002-2003, αν θυμάμαι καλά, υπάρχουν κάποιες εκθέσεις για τις συνέπειες των αξιολογήσεων αυτών. Καλό θα ήταν αν υπήρχαν τέτοιες μελέτες να εξετάζουμε περισσότερο την ποιοτική συνιστόσα ως παράμετρο. Μια τρίτη παρατήρηση στις απαντήσεις, στις γραπτές ερωτήσεις, συμβαίνει το εξής. Είχαμε και το θέμα της ερώτησης υπαριθμών 5, το θέμα δηλαδή των παρατυπιών. Κάποιες χώρες στην διαδικασία ανάκτησης ε, κονδυλίων αχρεωστήτως καταβληθέντων ε, είναι πραγματικά πρέπει να πω ουραγοί και βρίσκονται πολύ πίσω, χολένων το Βέλγιο, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στου ελέγχου που έκανε όσον αφορά το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιταλία, ερώτησή μου, ποια αποτελέσματα από αυτού του ελέγχου ε, μπορούμε να ε, θεωρήσουμε ότι συνήχθησαν. Αναφέρεστε στην απάντηση σε αυτή την πτυχή. Όμω το αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων στο Βέλγιο, Ιταλία, Ελλάδα, τα αποτελέσματα θα έπρεπε να διατεθούν στα μέλη τη κοινοβουλευτική μα επιτροπή. Αυτή είναι η παρατήρησή μου. Ευχαριστώ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λέει η κυρία Ιβάνοβα. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Ήθελα να θέσω ένα ερώτημα που έθεσα και χθες Γιατί την αυξημένη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην κοινή συγχρηματοδότηση για τις ε, χώρες μέλη που αντιμετωπίζουν ε, οικονομικές δυσκολίες. Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής για το θέμα αυτό. Από τη στιγμή που το ποσοστό χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγαλώνει σε σχέση με το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής, αυτό δεν σημαίνει ότι θα αυξηθεί και η πιθανότητα των σφαλμάτων δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής για αυτό το θέμα. Άλλωστε οι χώρες που έχουν οικονομικές δυσχέρειες είναι και οι χώρες που παρουσιάζουν τα περισσότερα προβλήματα σε όλο αυτό το θέμα. Άρα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυξημένοι έλεγχοι σε αυτά τα κράτη-μέλη. Και πιστεύετε ότι τέτοιου είδους επιβραβεύσεις, γιατί ουσιαστικά επιβράβευση είναι όταν δεν κάνει κανείς σωστά τη δουλειά του. Δεν θα πρέπει να υπάρχει επιβράβευση για τις χώρες που δουλεύουν σωστά, έχουν σωστή δημοσιονομική πειθαρχία και πληρούν τα κριτήρια του Μάστριχτ. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, δεν έχω άλλους ομιλητές στον κατάλογο. Έχω όμως ένα ερώτημα να θέσω εγώ ο ίδιος. Ε, πέρα, ε, επι, επιπρόσθετα, σε σχέση και με το ερώτημα του κυρίου Κεμπράντη, για το ποιος πληρώνει τελικά. Θυμάμαι αμυδρά, δεν ξέρω αν ισχύει, αν ισχύει ακόμα, το ε, ειδικό τέλος, την ειδική εισφορά στην ε, Ιταλία την πληρώνουν οι αγρότες ή η κυβέρνηση. Εγώ θυμάμαι, νομίζω ότι πληρώνει η κυβέρνηση, αλλά μπορεί η Επιτροπή να απαντήσει συγκεκριμένα. Να δώσω το λόγο τώρα στο ελεγκτικό συνέδριο. Έχουμε δύο μέλη διαθέσιμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να απαντήσω στα ερωτήματα που τέθηκαν στο ελεκτικό συνέδριο, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον ε, κύριο εισηγητή, τα μέλη της Επιτροπής σας και όλους εσάς για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε ε, κατά τη διάρκεια εξέτασης ε, των αποτελεσμάτων για το έτος 2010. Να τονίσω το πιο σημαντικό συμπέρασμα που έχουμε εξάγει μετά τους ελέγχους για αυτή τη χρονιά. Και δεν είναι νέα παρατήρηση αυτή που θα ήθελα να κάνω. Για άλλη μια φορά είδαμε ότι οι κίνδυνοι είναι σημαντικοί, παραμένουν σημαντικοί ως προς το ε, τις συναλλαγές στο βαθμό που δεν λειτουργεί σωστά το σύστημα Άγιαξ. Πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί το σύστημα Άγιαξ ε, ως ο Ναι, έχουμε αναλάβει αυτή τη δουλειά και θα την προχωρήσουμε. Το λέω αυτό για να απαντήσω στο ερώτημα του κυρίου Στάς. Ως προς το ερώτημα του κυρίου Φέλνερ. Ένα δήμα χρησιμοποίησε το ελεκτικό συνέδριο για το 2010 για να ε, εξετάσει το σύνολο των σφαλμάτων για τους φυσικούς πόρους και καταλήξαμε στο ποσοστό του 2,3% είχαμε 238 συναλλαγές και σε αυτές τις 238 είχαμε αρκετές συναλλαγές για άμεσες πληρωμές βάσει του Άγιαξ για τις οποίες μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι το ποσοτικοποιημένο σφάλμα της τάξης του 5% ήταν ελεύθερο από το ουσιαστικό σφάλμα, δεν είχε δηλαδή ουσιαστικό σφάλμα και κατά τα λοιπά ήμασταν κάτω από το κατόφλιο του 2%. Μιλάμε για 30,7 ε, δις και διατηρούμε όλα αυτά τα στοιχεία, τα έχουμε. Το ελεγκτικό συνέδριο, ωστόσο, για τα υπόλοιπα δεν μπορούσε να, ε, συμπεραίνει, να συμπεράνει ότι ε, τα υπόλοιπα, ε, για τα υπόλοιπα ήμασταν κάτω από το 2%. Είναι, δεν είναι συμπέρασμα της Επιτροπής αυτό, όχι του ελεγκτικού συνεδρίου. Για την επόμενη χρονιά τώρα, για το 2011, το ελεγκτικό συνέδριο αποφάσισε να έχει δύο διαφορετικά δείγματα. Ένα για το πρώτο πυλώνα και ένα για το δεύτερο πυλώνα. πολιτική για το περιβάλλον, θαλάσσιες υποθέσεις, αλία, υγεία, προστασία του καταναλωτή. Άρα θα έχουμε δύο δείγματα αναλόγως με το εκάστοτε ταμείο και έτσι θα έχουμε πιο ειδική διακρύβωση της κατάστασης. Πιστεύω κύριε Φέλνερ ότι του χρόνου θα είστε περισσότερο ικανοποιημένος με τα συμπεράσματά μας. Η υπόθεση στην οποία αναφερθήκατε ε, είχε συμπεριληφθεί στο δείγμα μας και το έχουμε συζητήσει το θέμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το λέμε και στην ετήσια έκθεση μας, όπου εμένως δεν θα το επαναλάβω εδώ. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι έχοντας λάβει τα στοιχεία από τα κράτη-μέλη, έχουμε παραπέμψει την υπόθεση στην Όλαφ ο φορέας εκμετάλλευσης είχε φτιάξει ένα σύστημα επαναπόλυσης προς τα καρατιμέλη με μόνο στόχο να παρακάμψει την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έχουμε ενδείξει γι' αυτό. Είχε χρησιμοποιήσει έναν άλλο φορέα εκμετάλλευση μέσω άλλου κράτου μέλου, ο οποίο δεν λειτουργούσε ω ανεξάρτητο έμπορο, δεν είχε αναλάβει καθόλου ε, χρηματοπιστωτικούς κινδύνους και είχαμε κάνει διαβούλευση με διάφορα ε, ε, όργανα. Τελικά είδαμε ότι αυτές οι δύο εταιρικέ οντότητες αυτό που ήθελαν ήταν να παρακάμψουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να μην υπάρχει μια πλήρως ανεξάρτητη συναλλαγή με ανεξάρτητα όργανα. Θεωρεί λοιπόν το ελεκτικό συνέδριο ότι είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει μόνο συμμόρφωση με το τυπικό αλλά και με το ουσιώδες της διαδικασίας. Δηλαδή η ουσία πρέπει να, ε, ε, να είναι υπεράνω ε, της τυπικής συμμόρφωσης με το διατακτικό. Δεν θα, να, δεν θα πρέπει να υιοθετείτε μία απλουστευμένη ανάλυση των νομικών διατάξεων. Μιλούμε για μεταφορές αγαθών ε, με πάνω από 500 φορτηγά σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 ε, χιλιόμετρων. Εκεί δεν θα πρέπει να ε, συμμορφούνται κανείς μόνο με, τη, με τις τυπικές διαδικασίες αλλά και με την ουσία, το πνεύμα του νόμου. Είναι στοιχεία που είχαμε δει το 2009 και όπως είπε και ο κύριο Φέλνερ στην ειδική μας έκθεση για τις ε, ε, ενισχύσεις σε διατροφικά προϊόντα ε, στα πρόσωπα που χρήζουν βοήθειας, η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί θα πρέπει να διακοπεί για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Τέλος, θα ήθελα να πω το εξή: Ο Επίτροπος κ. Σιόλος αναφέρθηκε στην πρόταση μεταρρύθμισης ε, της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής πέρα από το 2013. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία ε, για το ελεκτικό συνέδριο ε, να συμβάλλει σε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα λοιπόν ε, να σας πω ότι εμείς προετοιμαζόμαστε για να εκδώσουμε γνωμοδότηση για τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις της Επιτροπής για την επόμενη χρονιά. Από ό,τι φαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πράγματι ενσωματώσει στην πρόταση τις ε, προηγούμενες συστάσεις, συστάσεις προηγούμενων ετών του ελεκτικού συνεδρίου, κάτι το οποίο μα χαροποιεί ιδιαιτέρω. Αναφέρομαι κυρίω στον ενεργό δραστήριο αγρότη που όντω ασκεί αυτή την επαγγελματική δραστηριότητα, ε, την βιολογική γεωργία και Όλα αυτά μα χαροποιούν ιδιαιτέρω. Να δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου, τον κύριο Κρέντερ. Ο πρόεδρο. Ένα σύντομο ερώτημα ε, προς εσά από τον κύριο Φέλνερ προς εσάς κυρία Λεβίσελα. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Φέλνερ. Μόλις έμαθα ότι αυτή η υπόθεση μεταφοράς βουτύρου από την Ιταλία ε, προς τη Γερμανία δεν είναι παράδειγμα κακοδιαχείρισης, είναι πλέον υπόθεση ε, την οποία έχει αναλάβει η Όλαφ. Μόλις το μάθαμε και αυτό. Πιστεύετε πράγματι δηλαδή ότι πρέπει να διακοπούν αυτές οι ενισχύσεις Μέχρι ότου ξεκαθαριστεί η υπόθεση και ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, ε, λάβει μέτρα υπέρ της διαφάνειας. Πότε αποφασίσατε να παραπέμψετε την υπόθεση στην Όλαφ. Μέχρι σήμερα το πρωί, πριν, την, ε, πριν το ξεκίνημα της συνεδρίασης, θεωρήσαμε ότι ήταν απλά ένα παράδειγμα προς όχι μια υπόθεση της Όλαφ, το μέλος του ελεκτικού συνεδρίου. Ναι, ε, περιμέναμε όλες αυτές τις επιστολές, τις απαντητικές από πλευράς Ιταλικών αρχών. Όταν ε, συλλέξαμε το σύνολο των στοιχείων, μετά είχαμε μια πλήρη εικόνα και αποφασίσαμε να παραπέμψουμε την υπόθεση στην Όλαφ. Ο κύριος Κρέντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, είπε ο κύριος Αλεβία Λενίσελα, όταν συντάξαμε την έκθεση αυτή, δεν, είχε, δεν είχαμε ακόμα παραπέμψει την ε, υπόθεση στην Όλαφ γιατί περιμέναμε απαντήσεις από πλευράς Ιταλίας και κάτω χωρών. Επομένως, ε, Τώρα τις έχουμε και τις, ε, την παραπέψαμε στην Όλαφ. Το συμπέρασμα του ελεκτικού συνεδρίου είναι σαφέστατο. Σημειώνεται παράβαση των ευρωπαϊκών κανόνων σε δύο επίπεδο. Καταρχάς, εικονικά είχε εισαχθεί το βούτυρο αυτό στην Ιταλία και μάλιστα ποτέ δεν έφτασε, δεν ξεπέρασε τα τελωνία. Δηλαδή είχε εισαχθεί μόνο επί χάρτου. Δεν, δεν είχε γίνει ουσιαστική ε, εισαγωγή. Ε, αυτά τα τεμάχια βουτύρου δεν έφτασαν ποτέ σε ιταλικό έδαφος. Και απαιτεί ο κανονισμός να γίνει όντως εισαγωγή του βουτύρου. Ε, ξέρετε οι ελεκτές ότι, ε, ξέρετε ότι οι ελεκτές ακολουθούν τον εξής κανόνα. Προτιμούν το πνεύμα και όχι το γράμμα του νόμου. Επομένως, το βούτυρο αυτό δεν εισήχθη ποτέ ως αντικείμενο και αυτό είναι παράβαση των ευρωπαϊκών κανόνων. Δεύτερον, δεν θα έπρεπε να είχε επαναποληθεί στην χώρη αγορά, δηλαδή τη γερμανική αγορά και ε, τελικά επαναπολύθη. Δεύτερη παράβαση των κανόνων. και μάλιστα δεν πωλήθηκε στη γερμανική αγορά από τον Ιταλό εισαγωγέα, αλλά από έναν Ολλανδό εισαγωγέα. Αυτός ο Ολλανδός εισαγωγέας ήταν ένας πράκτορας του Ιταλού, δηλαδή ένας μεσίτης που είχε κάνει αυτή την προσφορά. Θα έπρεπε λοιπόν να είχε εισαχθεί στην Ιταλία, δεν θα έπρεπε να είχε επαναπολυθεί στη Γερμανία. Αυτά τα δύο στοιχεία δεν έχουν ε, εφαρμοστεί, επομένως ε, υπάρχει σημειώνεται παράβαση των ευρωπαϊκών ε, κανόνων κατά την άποψη του ελεκτικού συνεδρίου. Έξω και παραπέψαμε το θέμα στην όλα. Κάνετε διάφορε παρατηρήσει για την ανάπτυξη τη υπαίθρου. Σα εκπλήσει το γεγονό ότι έχουμε τόσο πολλά σφάλματα στο δεύτερο πυλώνα σε σχέση με τον πρώτο πυλώνα. Γιατί τα τη ανάπτυξη τη υπαίθρου εντάσσονται στο δεύτερο πυλώνα. Είναι σωστό αυτό, είναι αληθέ. Θα έχετε παρατηρήσει ότι το ε, ελεκτικό συνέδριο εντόπισε ποσοστό σφάλματος της τάξης του 0,7%. Αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 3,17. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις πολιτικές που αφορούν στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Το μέγεθος ε, των σφαλμάτων δηλαδή είναι ακόμα πιο σημαντικό, είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτό που ε, αναφέρετε εσείς. Πολύ ψηλό δηλαδή. Γιατί σε γενικέ γραμμέ μπορεί κανεί να δώσει μια εύκολη εξήγηση. Όσο περισσότερο μπαίνει στι λεπτομέρειε, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η εξήγηση. Σε γενικέ γραμμέ όμω μπορώ να πω το εξή. Έχουμε από τη μία πλευρά ένα απλό σύστημα, τον πρώτο πυλώνα. Χ εκτάρια, ε, άρα δικαιούται κανείς χι ε, άμεση ενίσχυση, ενιαία ενίσχυση, κάνει τον πολλαπλασιασμό και βρίσκει το νούμερο που θα πάρει. Είναι ένα απλό σύστημα αυτό να γίνεται εύκολα η διαχείρισή του. Στην ανάπτυξη της υπαίθρου, ε, στο δεύτερο πυλώνα, υπησέρχονται εκεί διάφορες ομορφές παρέμβασης. Παρέμβασης που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη υποδομών, με το περιβάλλον, με το γεωργικό περιβάλλον, με τα δάση, με πολλά και διαφορετικά πράγματα. Επομένως, σε ένα πλαίσιο όπου η νομοθεσία είναι πραγματικά πολύ περίπλοκη και οι στόχοι είναι πολύ πιο ε, πολύ και ποικίλοι, τότε εκεί καταλαβαίνετε ότι προκύπτουν πολύ πιο πολλές ευκαιρίες και περιπτώσεις για σφάλματα. Εξού και έχουμε αυξημένο ποσοστό σφαλμάτων ε, στα θέματα που άπτονται της ανάπτυξης υπαίθρου και εξού και πρόκειται να έχουμε αυξημένο ποσοστό σφαλμάτων για τα θέματα αυτά για περισσότερο χρόνο, σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Εάν θα βελτιωθεί η κατάσταση σε αυτό το τομέα, αυτό θα εξαρτηθεί από μια πιο ενδελεχή εξέταση όλων αυτών των προγραμμάτων για την ανάπτυξη της υπαίθρου που εφαρμόζουν και υλοποιούν τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται χρόνος. Το σύστημα Ajax το έχουμε εδώ και πολλές δεκαετίες, το έχουμε βελτιώσει σε βάθος χρόνου ε, ε, από χρονιά σε χρονιά. Έχουμε φτάσει τώρα σε ένα εύλογο, σε ένα λογικό στάδιο σε αρκετά ολοκληρωμένο, όμως το IPL ε, έχουμε αρκετά σφάλματα ακόμα δυστυχώς. Η κατάσταση δηλαδή δεν είναι βελτιούμενη, όμως όντως είναι ένα τομέα που εκτίθεται ε, σε περισσότερα σφάλματα. Ο κίνδυνος σφαλμάτων είναι αυξημένος. Και ένα τελευταίο σχόλιο για τις ε, τριμερείς συσκέψεις. Το ελεκτικό συνέδριο δεν είναι υπέρ των ε, τριμερών συσκέψεων και ο λόγος είναι ο εξής. Εμείς ελέγχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η, οποία έχει και την ε, τελική ευθύνη για τη διαχείριση του κοινοτικού ε, προϋπολογισμού. Ο ελεγχόμενος είναι η Επιτροπή. Το ελεκτικό συνέδριο δηλαδή ελέγχει την Επιτροπή και όχι τα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή παρουσιάζει τον προπολογισμό, τον ε, διαχειρίζεται και εμείς δίνουμε σε εσά μια γνωμοδότηση για τον τρόπο με τον οποίο έχει εκτελεστεί ο προπολογισμό. Σε τελική ανάλυση δηλαδή συνομιλητής μας είναι η Επιτροπή και αυτό κάνουμε. Γι' αυτό και είναι διμερής η στις σκέψεις μας, στις συνεδριάσεις μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως και χρειαζόμαστε τα κράτη-μέλη και μάλιστα στην πραγματικότητα ε, βασιζόμαστε στη βοήθεια όλων των κρατών μελών. Τους γράφουμε, τα χρειαζόμαστε, λαμβάνουμε γραπτές απαντήσεις από τα κράτη-μέλη και αξιοποιούμε όλες τις πληροφορίες που μας δίνουν. Ωστόσο, όταν έχει μετρηθεί εσφαλμένα ένα συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, για παράδειγμα, αυτό δεν θα βελτιωθεί. Η μέτρηση δεν θα βελτιωθεί ε, με το να υπάρχει εκπρόσωπος ε, των κρατών μελών ή του Συμβουλίου στην ε, σύσκεψη και να γίνει τριμερής η σύσκεψη αντί για διμερής. Δηλαδή, δεν, δεν θα διορθωθεί αντί για 2,9 εκτάρια να γραφεί το σωστό που είναι 2,1 εκτάρια. Το κράτος μέλος έχει απαντήσει γραπτός για το θέμα αυτό. Δεν καταλαβαίνω ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία της φυσικής παρουσίας ενός εκπρόσωπου του κράτους μέλους σε αυτή την συνεδρίαση. Και αν επανέλθουμε στην υπόθεση του Βουτύρου, τότε θα έπρεπε να έχουμε τέτραμερη σύσκεψη με την Επιτροπή, τη Γερμανία, την Ιταλία, τις κάτω χώρες και το ελεκτικό συνεδρίο, δηλαδή ε, σύσκεψη με ε, διαφορετικά, μεταξύ πέντε διαφορετικών μερών τελικά το, το ελεγκτικό συνέδριο θα εξάγει το συμπέρασμα. Αυτό είναι το καθήκον του. Και ε, το να υπάρχει και το να οργανωθεί διμερής, τριμερής, τετραμερής ή πενταμερής ε, συνεδρίαση δεν θα αλλάξει καθόλου την ε, κατάσταση. Σκοπός του ελεκτικού συνεδρίου είναι να έχει τη δυνατότητα να βλέπει την κατάσταση ξεκάθαρα ποια είναι τα γεγονότα. Ε, δεν έχει μεγάλη σημασία ο αριθμός ε, των παριστάμενων γύρω από τον ε, τραπέζι των, της σύσκεψης αυτής. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω το μεγαλύτερο δυνατό σταθμό, σταθμό της απαντήσεις και τα σχόλια. Είναι να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου αναγνωρίζω και το είπα και στην παρέμβασή μου ότι αν μιλούμε για ποσοστό λάθους ε, υψηλό, εάν θέλετε στην ΚΑΠ, μιλούμε για την ε, ανάπτυξη της υπαίθρου. Για τις άμεσες πληρωμές, όπως είπε το Ελληνικό Συνέδριο. Και ό,τι χειρίζεται το Θεογκά, η επαλήθευση του Ελεκτικού Συνεδρίου και στατιστικές δείχνουν ότι είμαστε κάτω από ποσοστό 2%. Τώρα, για την ανάπτυξη πέθρου. Εντόπισε στα μέτρα για το περιβάλλον το ελεκτικό συνέδριο πιο υψηλό ποσοστό σφάλματος, αλλά αυτό το ανέφερα επίσης στην παρέμβασή μου. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια, διότι η Επιτροπή έλαβε ήδη μέτρα εδώ και δύο χρόνια για να βελτιωθούν οι στατιστικές αφενός και για να διασαφινιστούν οι κανόνες ελέγχου ώστε να μειωθεί ο αριθμός των σφαλμάτων. Το 0,7 που ανέφερε ο κύριος Κρέτ, που δεν αναφέρθηκαν στο ποσοστό υλικού λάθος από το λεκτικό Συνέδριο αφορά κάποιες προκαταβολές που δόθηκαν στα κρατημένα. Δεν πρόκειται για αριθμητικό λάθος, διότι όντως πρόκειται για χρήματα τα οποία δόθηκαν και δαπανήθηκαν και εκεί ο έλεγχος έγινε όπως γίνεται και για τα υπόλοιπα χρήματα που καταβάλλονται. Ακόμη λοιπόν και έτσι το ποσοστό σφάλματος για την ανάπτυξη πέθρου μειώθηκε, αλλά και πάλι και εδώ φτάνουμε σε ένα επίπεδο από το οποίο, όπως ανέφερα και πέρσι, εξαιτία του γεγονότος ότι είναι ειδικά τα μέτρα που δίδονται για την περιφερειακή ανάπτυξη, που έχουν και πολιτικό στόχο, πράγμα που τα δύο θεσμικά όργανα δέχθηκαν, να μπορέσουμε να χειριστούμε οι ιδιάζοντα προβλήματα ε, αναπεριφέρεια. Δεν μπορούμε να πλουστεύσουμε περαιτέρω τα μέτρο, διότι δεν θα μπορέσουμε έτσι να υλοποιήσουμε τον πολιτικό στόχο που θέλουμε. Πρέπει λοιπόν δεχτούμε αυτό το ποσοστό πολυπλοκότητας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας αφάσεις λαμβάνοντας υπόψη τις διατερότητες των διαφόρων περιοχών. Αυτός είναι ο στόχος λοιπόν, να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε τους ε, ε, αγρότες να εφαρμόσουν κάποιες αγροτικές πρακτικές για την βιοπικιλότητα, για την ποιότητα του εδάφους, για το υδάτινους πόρους κτλ. Για την επόμενη όμως περίοδο προγραμματισμού, όπως έλεγα και προηγουμένως, ήδη λάβαμε μέρα, μέτρα ώστε να διευκολύνουμε τα πράγματα όσον αφορά τους ελέγχους, όσον αφορά τον ορισμό των μέτρων, όσον αφορά τους δείκτες για να μετρήσουμε και όσον αφορά το σύστημα EAX, το οποίο θα μας επιτρέψει να κάνουμε καλύτερο έλεγχο όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Συνεχίζουμε λοιπόν τις προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση. Κυρία Φέλνερ, ρωτήσατε γιατί υπάρχουν διαφορές μεταξύ διαρθρωτικών ταμείων και ταμείο ε, ανάπτυξης υπέθρο όσον αφορά το ποσοστό σφαλμάτων. Η απάντηση είναι ότι προσπαθήσαμε να αφηγραμμίσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα μέτρα τα πρώτα, ο, με τρόπο που να μπορούν να ελέγχονται από την ΆΙΕΞ που έχει βάσεις δεδομένων που παρά τις ε, αδυναμίες που έχουν δεν επηρεάζουν τις δαπάνες. Και όπως είπε ο κύριος Κρέτε, έχουμε ε, αγροτεμάχια στο σύνολο της Ένωσης περίπου της τάξεως των ε, Δεκάδες χιλιάδων εκατομμυρίων και γι' αυτό εμφανίζονται μικροσφάλες. Όταν γίνονται επιτόπου έλεγχοι ε, και τους διασταυρώνουμε με άλλους ελέγχους που γίνονται, κάνουμε επαληθεύσεις και διορθώνουμε λάθη χωρίς αυτό να έχει στα διάφορα κονδύλια επιπτώσεις. Επίσης για την ανάπτυξη της υπαίθρου που χειρίζεται η ΕΚΣ γίνονται επίσης οι έλεγχοι, οι πράγμα που μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε από το ένα χρόνο στον άλλο που υπάρχουν ε, σφάλματα και να κάνουμε, βλάβουμε διορθωτικά μέτρα οικονομικά. Διότι όταν έχουμε συστημικά λάθη μπορούμε να προβλέψουμε ε, τρόπους βελτίωσης του ελέγχου ακόμη και στο δεύτερο πυλώνα. Το σύστημα ελέγχου και τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται για να βελτιωθεί το σύστημα ελέγχου, αλλά συγχρόνως οι διορθωτικοί λογαριασμοί που γίνονται μας επιτρέπουν από τον ένα χρόνο στον άλλο να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν προβλήματα. Και εδώ και κάποια χρόνια επίσης έχουμε αυτή την συμπληρωματική ασφάλεια που μας παρέχουν οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης στο σύνολο του προϋπολογισμού στον πρώτο πυλώνα και στον προπολογισμό που διατίθεται για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτοί λοιπόν οι κανόνες μας κάνουν να μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα το τι γίνεται από το ένα χρόνο στον άλλο και να διορθώνουμε τα προβλήματα όταν εμφανίζονται και να μην περιμένουμε να χρονίσουν. Όσον αφορά την ανάκτηση. Και εδώ ανέφερα στην εισαγωγικές μου παρατηρήσεις ότι μετά από τις παρατηρήσεις που έκανε το ελεκτικό συνέδριο και τις συζητήσεις που είχαμε πέρσι, την έκθεση του κυρίου Χατζημαρκάκη, ενθαρρύνουμε το σύστημα να συνεχίσει με τον τρόπο που λειτουργήσει, οπότε να έχουμε καλύτερες ανακτήσεις. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι την παρακολούθηση του τι γίνεται εκ των υστέρων και βλέπουμε ότι το ποσοστό των ανακτήσεων αυξήθηκε. Έχουμε ένα σύστημα τώρα που είναι της τάξης του 50-50. Σε περίοδο 4 ή 8 ετών, τα κράτη-μέλη τα οποία δεν ανέκτησαν το 50% των ποσών μας λέτε ότι καλείται να πληρώσει δύο φορές ο φορολογούμενος. Εμείς όμως Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη, είναι 27. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Αλλά βλέπουμε το, με το 50-50 ενθαρρύνονται τα κράτη-μέλη να ανακτήσουν τα χρήματα από το Δεν δεδομένου ότι η κατάσταση βελτιώθηκε πάρα πολύ. Είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία τώρα το ποσοστό ανάκτηση το πρώτο έτος ξεπερνάει το 25%. Ενώ βλέπουμε ότι προηγουμένως σε περίοδο πενταετή Είχαμε ανάκτηση 20% ενώ τώρα τα 4 χρόνια βλέπουμε να ξεπερνιέται και το 50%. Γι' αυτό τώρα περάσαμε σε αυτό το σύστημα και θέλουμε να φτάσουμε στο τέλος, στο τέλος περίοδου ανάκτηση ποσοστό 100%. Και αν κάποιο κράτος δεν έχει ανακτήσει όλο το σωστό, μπορεί να παρέμβει η Επιτροπή ώστε να ανακτήσει τελικά το 100% των οφειλούμενων ποσών. Τώρα, γιατί υπάρχουν διαφορές μεταξύ αυτού το οποίο υπολογίζουν τα κράτη-μέλη ως διόρθωση που πρέπει να εφαρμοστεί για την ανάκτηση και αυτό το διαπιστώνεται από την Επιτροπή. Και αναφέρεται την περίπτωση της Ελλάδας. Αυτό συμβαίνει διότι εκτός από αυτό το οποίο ανοιχνεύουν ως φάλμα στον τελικό δικαιούχο το κράτο μέλος και εμείς ανοιχνεύουμε κάποια συστημικά σφάλματα και εκεί εφαρμόζουμε το διορθωτικό ε, δίκτυο όπως στην περίπτωση της Ελλάδας. Αυτό έγινε, διότι διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν στη βάση δεδομένων και στο σύστημα IPS κάποια λάθη και γι' αυτό κάναμε κάποιες ε, ε, οικονομικές διορθώσεις ώστε τα λάθη αυτά να μην επαναληφθούν. Στο σύστημα που υπήρχε στην Ελλάδα δεν μπορούσαν καταρχά να ανοιχτευτούν αυτά τα λάθη. Όταν έγινε όμω οικονομικό έλεγχο, διαπιστώθηκαν. Γι' αυτό υπάρχουν διαφορέ μεταξύ αυτού που διαπιστώνουν τα κράτη-μέλη και αυτών το οποίο διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι, εάν εμεί εντοπίσουμε ένα σφάλμα σημαντικό στην ποιότητα της βάσης δεδομένων των αγροκτημάτων και των ελέγχων που γίνονται επί τόπου, θεωρούμε ότι η χρησιμοποίηση ε, των κοινοτικών κονδυλίων επηρεάζεται, τα ανακτούμε και χρειάζεται να διορθώσει τη βάση δεδομένων το κρατομέλων. Επίσης, μου είπατε να κάνω μια σύγκριση σχέση με το διορθωτικό ε, σύστημα. Υπάρχει αυτό το κίνητρο με αυτό το σύστημα. Πρέπει να πω ότι πολλές φορές δεν χρειάστηκε να μπλοκαριστούν οι πληρωμές, διότι το μπλοκάρισμα είναι συγκυριακό πρόβλημα. Προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα συγκυριακά. Δεν γίνεται η πληρωμή, αλλά αν παραμείνει το σφάλμα στο σύστημα, θα παραμείνει ακόμη και όταν καταβληθούν τα χρήματα. Οι οικονομικέ λοιπόν διορθώσει είναι κάτι που επιτρέπει στα διάφορα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τα συστήματά τους. Και αναφέρουμε την περίπτωση της Ελλάδας, της Ρωμανίας, της Βουλγαρίας και τώρα βλέπουμε μετά από του οικονομικούς ελέγχους ότι η κατάσταση βελτιώθηκε σε αυτέ τι χώρε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την ανάκτηση. Επίσης ανέφερα τα μέτρα με το πέρασμα σωστή σύστημα από το 50-50 στο 100% αλλά διευκρινίσαμε και περισσότερο την κατάσταση που πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν, δηλαδή να καταγράφουν το ακριβώ γίνεται και να παρακολουθούν εκ το σύνεγγυ τις ε, εξελίξεις. Και πολλές φορές εδώ ε, έχουμε απέναντί μας την εθνική νομοθεσία, διότι πρέπει να περιμένουμε την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και τις αποφάσεις των δικαστηρίων πριν να μπορέσουμε εξονόμετρα της Επιτρόπης να ενεργήσουμε για να ανακτήσουμε κάποια ποσά. Γι' αυτό η ενιοποίηση και τυποποίηση των συστημάτων έχει και τα όρια της. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε παντού τις ίδιες αρχές και κανόνες, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε δηλαδή να παρέμβουμε εκεί που πρέπει η δικαιοσύνη να βρει τη λύση. Στην Ισπανία, στην Ιταλία, Φερρυπίν. Και χρονίζουν πολλές φορές οι αποφάσεις. Πρέπει όμως να τις περιμένουμε. Ακόμη και πριν εφαρμοστεί η εθνική νομοθεσία σε περίπτωση ε, στάσεις πληρωμών. Βεβαίως λέγω ότι υπάρχουν και περιορισμοί σε κάθε εθνική νομοθεσία και δεν υπάρχει εδώ πλήρης ευθυγράμμιση. Τώρα σε όρες της αναφορά το βούτυρο. Εδώ και για να επανέλθουμε το θέμα των τριμερών συναντήσεων. Εγώ δεν ζήτησα να έχουμε τριμερείς συναντήσεις για περιπτώσεις οι οποίες είναι ε, προφανείς. Πολλές φορές έχουμε μία νομοθετική ερμηνεία σε κάποιες περιπτώσεις, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει την νομοθεσία που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και βάσει αυτής της νομοθεσία και των κανονισμών λαμβάνουμε αποφάσεις αν, μπορούμε, αν πρέπει να ανακτήσουμε χρήματα, αν έχουμε να κάνουμε αριθμητικό λάθος ή έχουμε περίπτωση απάτης. Και δεδομένου μοιραζόμαστε τη διαχείριση εάν η Επιτροπή και το κράτο μέρος αποφασίσουν να κάνουν την ε, τριμερή συνάντηση, μπορούμε να διευκρινίσουμε τα θέματα παρερμηνίας πιο εύκολα. Αυτός ο μηχανισμός εφαρμόζεται όμως από το ελεκτικό συνέδριο στην περίπτωση των διαρθρωτικών ταμείων. Και για τον δεύτερο πυλώνα, για την ανάπτυξη τη ημέθρου, υπάρχουν ε, σημεία που ομοιάζουν με αυτή την κατάσταση. Εάν λοιπόν τα επιχειρήματα του κυρίου Κρετέ ίσχυαν και για την ΚΑΠ, γιατί να μην είναι για την πολιτική συνοχής. Ζητήσαμε απλώ να χειρίζεται το θέμα αυτό με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα θέματα των διαρθρωτικών ταμείων το ελεκτικό συνέδριο. Όχι γενικά, αλλά όταν υπάρχει ανάγκη να γίνει γρηγορότερα και καλύτερα διευκρίνηση μιας κατάστασης η οποία δημιουργεί ερωτηματικά. Τώρα, στην περίπτωση του βουτήρου η θέση της Επιτροπής ήταν ότι δεν υπήρξε παραβίαση των κανονισμών τα κράτη-μέλη που ενέχονται σε αυτήν την υπόθεση και οι διάφοροι φορείς σεβάστηκαν την ομοθεσία και γι' αυτό το λόγο δεν θεωρήσαμε εμείς ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να ανακτηθούν. Ίσως υπάρχουν αδυναμίες στους κανονισμούς. Δηλαδή, τι κάνουμε σε περίπτωση που έχουμε μεγάλα αποθέματα. Και τα αποθέματα εν μέρη τα πολλούμε. Δεν τα δίδουμε μόνο στους ενδεείς. Τα πολλούμε για να χρηματοδοτούν τα προγράμματα. Ίσως θα πρέπει όλος όλος μηχανισμός να βελτιωθεί. Και από το 2014 ούτως ή άλλως δεν θα εφαρμόζεται πλέον αυτός ο μηχανισμός και για το 2012 και 2013 θα τον εφαρμόσουμε διότι δεν έχουμε πλέον ε, αποθέματα που θα μπουν στην παρέμβαση. Αλλά για το 2009 αυτός ο κανόνας να μην διατεθούν στις ε, ε, κάποιες ε, ποσότητες στις εθνικές αγορές ήταν ειδικά για το 2009, ώστε το βούτυρο που οποίο απεσύρθη από την εσωτερική αγορά να φτάσει στην ίδια αγορά τη στιγμή που εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Οι φορείς όμως οι διάφοροι σεβάστηκαν τους κανόνες και την νομοθεσία. Αυτή είναι η γνωμοδότηση της Επιτροπής και η άποψή μας, δεδομένου ότι το βούτυρο από τη Γερμανία χρηματοδότησε το πρόγραμμα των πλέον ενδυνών στην Ιταλία και ο Ιταλός φορέας για να έχει χρήματα και να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα πώλησε το βούτυρο αλλά από τη στιγμή που πωλήθηκε το βούτυρο αυτό κυκλοφόρησε στην Ιταλική αγορά. Δεν μπορούμε, οπουδήποτε, δεν μπορούμε να το εμποδίσουμε να πάει στην Ολλανδία ή στη Γερμανία. Πρόκειται για τον κανόνα της εσωτερικής αγοράς. Και ο στόχο ήταν να χρηματοδοτήσουμε το πρόγραμμα της πλέον ενδεής. Δεύτερον, το βούτυρο, να μην φτάσει στη στιγμή που είχαμε την περίοδο κρίσης στις αγορές που είχαν το πρόβλημα. Οι στόχοι αυτοί επιτεύθηκαν και οι κανόνες ικανοποιήθηκαν. Τώρα, το ότι είχε δυναμία στην νομοθεσία, αυτό είναι κάτι το οποίο πιστώσαμε και σε άλλε περιπτώσει. Και είναι απαραίτητο να γίνουν βελτιώσει και θα γίνουν δεδομένου ότι το πρόγραμμα θα, θα αλλάξει εντελώς βάσει της νομοθεσίας. Αυτή είναι η ερμηνεία μας για την περίπτωση αυτή. Τώρα, όσον αφορά το πρασίνισμα. Κύριε Φέλνερ, το αναφέρετε το θέμα. Είπατε ότι είναι πολύπλοκο. Μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω, αλλά το θέμα αυτό θα το συζητήσουμε όταν συζητήσουμε περαιτέρω τι νομοθετικέ προτάσει, ότι τα μέτρα που προτείναμε για το πρασίνισμα είναι τα πιο απλά. Θα χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο μηχανισμό ελέγχου επιτόπου με αυτόν που έχουμε τώρα για τι άμεσε πληρωμέ και ο έλεγχο θα γίνεται κατά τη διάρκεια τη ίδια περίοδου. Δηλαδή προσπαθήσαμε να μειώσουμε στο μέγιστο δυνατό την πολυπλοκότητα του συστήματος, αλλά πρέπει να σας πω ότι ξέρουμε ότι πρέπει να χειριζόμαστε σωστά τα χρήματα ευρωπαϊκά, αλλά πρέπει να καταλήγουμε και σε αποτελέσματα. Και ο κύριο Τάσα τόνισε το κατά πόσον θα πρέπει να είναι αποτελεσματική η πολιτική ποιότητα που θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε μελέτε αξιολόγηση και γίνονται όχι μόνο κάθε φορά που γίνεται επιτόπου έλεγχος, αλλά οι αξιολογήσει γίνονται κάθε φορά που προετοιμάζουμε μία μεταρρύθμιση. Όταν προσπαθούμε δηλαδή να βελτιώσουμε το σύστημα υποστήριξης προς τους αγρότες και να αποφευθούν καταστάσεις όπως αυτές που αναφέρατε. Τώρα, στην περίπτωση του βαμβακιού. Έχουμε μία ειδική κατάσταση. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ειδικό προϊόν. Αλλά στο σύστημα άμεσων πληρωμών έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι διαχωρισμένο. Δεν δίδονται οι πληρωμές ανά εκτάριο, αλλά για τα εισοδήματα του αγρότου. Και έτσι έχει αρκετά μεγάλο περιθώριο ο αγρότης για να ε, μπορέσει να διαπραγματευτεί το ενίκιο των γεών που ενοικιάζει από τον γεωκτήμονα. Και επαναλαμβάνω, δεν αφορούν το εκτάριο ετησίως, αλλά αυτόν ο οποίος νοικιάζει τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Και εδώ έγιναν βελτιώσεις και με το σύστημα που προτείνουμε για μετά το 2014 στοχεύουμε πολύ καλύτερα τις διάφορες ε, επιδοτήσεις που δίδουμε για τους νέους, για τις μειονεκτούσες περιοχές κτλ. ώστε να στοχεύουμε την υποστήριξη αυτή την οποία χορηγούμε καλύτερα και να μην υπάρχει μεγάλο περιθώριο σφάλματος όπως αναφέρατε εσείς ή παρερμηνίας. Τώρα σαν αφορά το θέμα της ανάκτησης, νομίζω ότι το ανέφερα, τα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος είπα ότι είναι πιο πολύπλοκα. Αλλά και πάλι βλέπουμε ότι υπάρχουν βελτιώσεις. Η ανάκτηση, κύριε Στάς, εξήγησε γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ αυτό το οποίο διαπιστώνουν τα κρατημέλη και ποσού το οποίο εμείς ανακτούμε όσον αφορά τη διαφάνεια. Ευχαριστώ που αναφέρατε το θέμα. Πρέπει να σας πω ότι για μένα είναι ένα θέμα πρωταρχικής σημασίας, διότι θέλω τον φορολογούμενο να δίδω την δυνατότητα να ξέρει πού πηγαίνουν τα χρήματά του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει αυτή τη στιγμή νέα νομοθεσία, λαμβάνοντα υπόψη τι παρατηρήσει που έκανε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επί αυτού του θέματος για την προσήτηση της ειδικής ζωής των φυσικών προσώπων και θα βρούμε κάποιο μηχανισμό ώστε οι μεγάλοι δικαιούχοι και οι επιχειρήσεις επίσης να υποφελούνται από αυτή την διαφάνεια και θα επανέλθουμε με νομοθετική πρόταση. Κυρία Εβάνοβα, για την συγχρηματοδότηση των χωρών που έχουν δυσκολία. Το γεγονός ότι αυξάνεται η συγχρηματοδότηση δεν επηρεάζει το ποσό των ελέγχων. Μόνο το επίπεδο συγχρηματοδότησης θα φτάνει. όχι το τελικό ποσό. Και οι έλεγχοι που κάνουμε είναι οι ίδιοι με το παρελθόν. Δεν συμβαίνει ότι επειδή δίδουμε περισσότερο ποσοστό ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερους ελέγχους ή διαφορετικούς, γιατί πάντα ε, έχουμε τον ίδιο αριθμό ελέγχων τους οποίους κάνουμε δειγματοληπτικά. Πάντα ότι δεν παίρνουμε πάντα τις χώρες που λειτουργούν τον καλύτερο τρόπο, αλλά βεβαίως η χρηματοδότηση δεν αυξάνεται. Για τις χώρες που έχουν κακή διαχείριση, αλλά για τις χώρες που έχουν οικονομικά πρόβλημα. Η Ελλάδα είχε οικονομικά προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι κάναμε λιγότερους ελέγχους. Η ποιότητα του ελέγχου και το επίπεδο συγχρηματοδότησης μπορεί να είναι διαφορετικό. Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε λιγότερο απαιτητικοί με τις χώρες αυτές. Αυτό απεδείχθη και με τη Βουλγαρία και με την Ρουμανία και με την Ελλάδα καθώς και με τις άλλες χώρες οι οποίες άλλαξαν τα πράγματα. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις που κάνατε. Τα ποσοστά ε, γάλα και το τέλος καταβάλλεται ε, για το γάλα στην Ιταλία. Από ποιον καταβάλλεται. Σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή ήδη ζήτησε από την Ιταλία να προχωρήσει στην ανάκτηση σύμφωνα με τον κανόνα 50-50. Παρακολουθούμε όμω εκ του σύνεγγυ όλη τη διαδικασία, τη νομική, στην Ιταλία, ώστε να μπορέσει να ανακτήσει η Ιταλία εκ μέρου των παραγωγών τα χρήματα. Ήδη έχουν γίνει κάποιες ανακτήσεις, αλλά υπάρχουν ακόμη ε, ε, διαδικασίε που εκκρεμούν στη δικαιοσύνη, Όσον ακόμη δεν έχουν λοιπόν οι εθνικέ αρχέ διευκρινίσει ποιο πρέπει να πληρώσει και τι ποσοστά, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω. Αλλά παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ με τις Ιταλικές αρχές την εξέλιξη των προμάτων και είναι και η περίπτωση της Ισπανίας. Πολλές φορές ε, τρενάρει η δικαιοσύνη όσον αφορά την οριστική τη απόφαση. Και αν δεν έχουμε την απόφαση των δικαστηρίων, εμείς κατά την απόψή μας δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο, αλλά παρακολουθούμε τι εξελίξει. Ευχαριστώ κυρία Γκρέσλερ για το θέμα των ποσοστώσεων γάλακτος και τις απάτες. Θα μπορούσαμε να έχουμε κατάλογο όλων των περιπτώσεων απάτης ή προβλημάτων σχέση με τα ποσοστά γάλακτος στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι και εγώ επισήμανα μία περίπτωση στην Ισπανία, εσύ κάποια στην περίπτωση στην Ιταλία. Νομίζω λοιπόν ότι για να παρακολουθούμε την εξέλιξη των καταστάσεων, καλό θα ήταν να έχουμε έναν κατάλογο. Κύριε Επίτροπε, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, βεβαίω. Μπορεί, μπορεί. Θα σας δώσουμε όλα τα στοιχεία, αλλά και πάλι λέγω ότι μπορούμε να σας πούμε πώς έχει κατάσταση σήμερα, τι πώς έχουμε ανακτήσει, τι μπορούμε να ανακτήσουμε και ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά την ανάλυση ε, που κάνουμε εμείς για, σε κάθε περίπτωση και σε τι στάδιο βρίσκονται τα πράγματα σχέση με τις αποφάσεις δικαιοσύνη. Κάποιο άλλο Ευρωβουλευτή που θα ήθελε να σχολιάσει επί των τοποθήσεων του συνεδρίου ή τη Επιτροπή. Εσεί φυσικά κύριε Φέρνερ, αλλά ρώτησα άλλα μέλη. Δεν υπάρχουν άλλοι. Ο κύριος Φέρνερ τώρα για τις, τα συμπεράσματά σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομο. Νομίζω είχαμε μια πολύ καλή παρέμβαση και πολύ καλές συζητήσεις ε, για όλα τα θέματα. Ήταν πολύ καλό να μάθει κανείς, να μάθουμε περισσότερα για την ε, υλοποίηση, πώς ε, οι κυρώσεις προχωρούν, να υπάρχουν οι διαφοροποίησεις και οι διαφορές, όχι μόνο σε αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τις διαφορές μεταξύ ιδίων τομέων, ας το αποκαλέσω έτσι θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε ξανά το θέμα του βουτύρου νομίζω ούτως ή άλλως στο μέλλον. Πρέπει επίσης να προσθέσω ότι ίσως αυτό από την, ε, το θέμα των ε, τριμερών ε, συναντήσεων και μη τριμερών συναντήσεων άκουσα ευδιάκριτα αυτό το οποίο παρετήρησε το Ελεκτικό συνέδριο για τις διμερείς συναντήσεις αντί τριμερείς ή Άλλε συναφείς. Πρέπει να ομολογήσω ότι τίνω να συμφωνήσω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πραγματικά αν ε, περιτεύει πλέον να ασχολείται κανείς με αυτά τα θέματα αν δεν υπάρχει η σωστή εξίσωση και φαίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ικανοποίηση. Όμως ίσως δεν είναι αναγκαστικά αυτή η λύση όπως αφελώς έγινε υπενιγμός για το βούτυρο π.χ. πιο πριν. Διότι διαβάζοντας την απάντηση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου σαφέστατα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι στην περίπτωση του βουτύρου δεν βλέπει κάποια βάση για ανάκτηση των ποσών αυτών ουσιαστικά. Κανονικά θα το κατανοούσα ότι όταν υπάρχει ένα θέμα σφάλματος ή όταν υπάρχει περίπτωση από την άλλη πλευρά απάτης, όμως το συνέδριο λέει ξεκάθαρα απάτη η Επιτροπή λέει συνεχίζεται η κανονική ως ε, ε, ήθιστε διαδικασία και νομίζω ότι ναι με το γράμμα του νόμου ε, ήταν κάτι το οποίο έγινε σεβαστό αλλά το γράμμα είναι αποδυναμωμένο το πνεύμα πρέπει να γίνεται σεβαστό αυτό αποκόμισα από την παρέμβαση του ελεγκτικού συνεδρίου όταν γίνεται προσπάθεια να παρακαμφθεί ακόμα και το γράμμα του νόμου, ε, τουλάχιστον θα πρέπει να συναγάγουμε τα σωστά συμπεράσματα, να μάθουμε κάτι παραπέρα. Και γι' αυτό θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε το θέμα του βούτυρου. Σε αυτή τη φάση θα ήθελα να μάθω κάτι περισσότερο επί της ουσίας για αυτή την περίπτωση και όχι να έχουμε ε, εκτενείς συζητήσεις μόνο για θέματα λεπτομέρειας ε, που δεν είναι τόσο ουσιώδη. Όπως είπα όμως ήταν καλή η θετική αυτή η συνεδρίαση και έχουμε τη βάση, τα θεμέλια για να προχωρήσουμε και να συναγάγουμε συμπεράσματα από αυτά. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν. Ε, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο από αυτά τα συμπεράσματα τα οποία διατυπώσατε. Ήταν πολύ καλά και όλοι συμμετείχαν, το Ελληνικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θετικό τρόπο. Και έτσι νομίζω εξαντλήσαμε το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ όλους σας. Avec ces deux types, ils sont ici ou non? Sorry? Yes, I think they are. Σε περίπτωση που κάποιος θα ήθελε να συνεχίσει τις συζητήσεις, παρακαλώ να βγει και να συζητήσει εκτός αίθουσας. Θα ήθελα να συνεχίσουμε με τις εργασίες μας, αν γίνεται, με το σημείο 7. And... Και θα ήθελα Παρακαλώ, καθίστε. Κύριε Σκούμπικ θα λάβει τον λόγο παρακαλώ από το ελεγκτικό συνέδριο για την εισαγωγή της ε, έκτακτης ειδική έκθεση ε, για το γάλα, για τα σχολεία και τα φρούτα στα σχολεία, αν είναι αποτελεσματικό αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, <clears throat> Κυρίε και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε έναν έλεγχο τη αποτελεσματικότητα των δύο αυτών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γάλα για τα σχολεία και τα φρούτα για τα σχολεία. Επιτρέψτε μου σύντομα να παρουσιάσω τα συμπεράσματα και τι συστάσει. Χρηματοδοτείται το γάλα εδώ και πάνω από 30 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με απλά λόγια επιτρέπει το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα σε ε, προσιτές μειωμένες τιμές ε, να είναι διαθέσιμα στους μαθητές. Και τώρα αν γάλα, τυρί, γιαούρτι προσφέρονται στους μαθητές ε, μέσα στο πλαίσιο του δεκατιανού τους στη σχολική καντίνα ή εκτός, αυτό είναι θέμα επιλογής που γίνεται από τα σχολεία. Κάθε ένα και όλα τα σχολεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Για τα φρούτα είναι καινούριο το πρόγραμμα. Ξεκίνησε το 2009. Έχει ειδικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την εθνική στρατηγική για τα φρούτα και την διανομή των φρούτων και των οπωρολαχανικών που είναι άνευ ε, καταβολής τέλους δωρεάν και γίνεται ε, κανονικά στα σχολεία πρέπει να ολοκληρώνεται να συμπληρώνεται με κάποιες παιδαγωγικές δραστηριότητες. Και τα δύο προγράμματα έχουν την ίδια βασική προσέγγιση, την διάθεση αυτών των προϊόντων στα σχολεία στους μαθητές, ώστε να επιτυγχάνονται οι ίδιοι κοινοί στόχοι και σκοποί, να, σταθεροποιηθεί, να σταθεροποιηθούν οι αγορές, αυτό είναι ο στόχος υπερσταθεροποίησης των αγορών και να προαχθεί η υγεία, να είναι καλύτερη για των μαθητών. Και οι δύο, τα δύο προγράμματα στοχεύουν στους δύο ίδιους στόχους για την διατήρηση και διασφάλιση και αύξηση των επιδοτούμενων προϊόντων αυτών στους νέους με τη διάθεση αυτών των προϊόντων στα σχολεία και μακροπρόθεσμα με την παιδαγωγική επιρροή που θα ασκηθεί με την εκπαίδευση όσον αφορά καλές τροφικές διατροφικές συνήθειες. Να υπογραμμίσω όσον αφορά την πρόσφατη φάση των φρούτων ο έλεγχος έγινε ακριβώς ε, για το γάλα όπου είχαμε ε, συγκρίσιμα στοιχεία ε, σχετικά βρίσκει το ελεγκτικό συνέδριο ότι το γάλα και μακροπρόθεσμα και βράχυπρόθεσμα ε, μικρή πίπτωση έχει. Μακροπρόθεσμα, βράχυπρόθεσμα δεν είναι πολύ αποτελεσματικό. Δεν είναι θελκτικό λόγω του χαμηλού επίπεδου ενίσχυσης ε, σε σχέση και με το γραφειοκρατικό βάρος που συνεπάγεται. Και επιπλέον υπάρχει η ιδιαίτερη δυσκολία να αποφύγουμε το βάρος της ε, ε, διανομής μέσω καντίνας, ε, μέσω κηλικίου σχολείων σε σχέση με τα τακτικά γεύματα. Στις περισσότερες δηλαδή περιπτώσεις τα προϊόντα για τα οποία καταβάλλεται η ενίσχυση στην, από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να είχαν συμπεριληφθεί και στα ε, γεύματα των καντίνων αυτών χωρίς ε, ακόμα και επιδότηση. Και βλέπουμε ότι δεν λαμβάνεται υπόψη ε, επαρκώς η επίτευξη των στόχων. Δεν υπάρχει συνάρτηση μεταξύ του παιδαγωγικού στόχου αυτών των προγραμμάτων και των επιδόσεων. Δεν γίνονται ιδιαίτερα ευδιάκριτα αυτά τα προγράμματα και δεν υπάρχουν άλλα παιδαγωγικά θα έλεγα κίνητρα ή μέτρα που να έχουν προαχθεί. Ας το δούμε σε βάθος χρόνου. Το 1999 σύστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Συμβούλιο ότι θα έπρεπε να καταργηθεί αυτό το πρόγραμμα διότι η αναλογία κόστους κόστους-οφέλους ε, δεν ήταν ε, θετική. Αποφασίστηκε να συνεχιστεί το πρόγραμμα και παρότι υπήρξε, υπήρξε ένας αριθμός ε, θετικών αλλαγών από το 1999 τα σημαντικά προβλήματα τα οποία σας παρουσίασα παραμένουν αν, χωρίς να έχουν επιλύθει. Από την άλλη πλευρά και θα ήθελα να το τονίσω, να το υπογραμμίσω αυτό, βρίσκουμε ότι οι περισσότερες αδυναμίες που εμείς οι ίδιοι διακριβώσαμε και εντοπίσαμε όσο αφορά το πρόγραμμα για το σχολικό γάλα σημειώθηκαν και τουλάχιστον εν μέρει ελήφθησαν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον προγραμματισμό των επισητιστικών αυτών προγραμμάτων. Σαν αποτέλεσμα, για, στο πρόγραμμα για το σχολικό γάλα έχουμε ένα τυποποιημένο πρότυπο διανομής, χωρίς ε, επιβάρυνση τελών και εκτός ε, καντίνων. Επίσης ε, συνοδευτικά παιδαγωγικά μέτρα έχουν ακολουθηθεί και ένα σημαντικό μέρος αυτού του προγράμματος θα έπρεπε και σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής να διασφαλίζει την ικανοποιητική, την επιτυχή εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Ενώ ακόμα είναι πρόημο να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτού του νέου προγράμματος, παρόλα αυτά φαίνεται ότι είναι πιθανότερο να επιτύχει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους όπως έχουν τεθεί. Και μια και είναι πολύ περιορισμένη η επίπτωση αυτού του προγράμματος, το μέλλον Δηλαδή, αν θα διασφαλιστεί ή όχι, θα πρέπει να εξαρτάται από όρους και προϋποθέσεις μεγάλων βαθέων μεταρρυθμίσεων που θα μπορούσαν πραγματικά μόνο αυτές να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες και τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν βασιζόμαστε στα εξή συμπεράσματα. Πρώτον, αν θέλουμε να έχει επίπτωση στον όγκο γάλακτος που καταναλώνεται στα σχολεία, η επιδότηση ανά λίτρο πρέπει να αυξηθεί σημαντικά σε ένα τέτοιο επίπεδο όπου το γάλα θα μπορεί να διανέμεται χωρίς επιβάρυνση οικονομική. Να τονίσω ότι αυτές οι συστάσεις δεν θα οδηγούσαν αυτόματα σε αύξηση των ε, κονδυλίων που δαπανάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αντίθετο, θα σήμαινε επικέντρωση κονδυλίων σε ένα στενό πλαίσιο του στοχοθετημένου πληθυσμού και θα καθορίζεται αυτός ο στοχοθετούμενος πληθυσμός από τις επισητιστικές ανάγκες. Δεύτερον, πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί η επιβάρυνση σε σχέση με τη διανομή από καντίνε και να διασφαλιστεί η μέγιστη, ο μέγιστο ευδιάκριτος χαρακτήρας, η ορατότητα του προγράμματος. Δεύτερον, τα δύο αυτά προγράμματα θα πρέπει να υιοθετήσουν και να προσαρμοστούν σε ένα πιο εναρμονισμένο, μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά μέτρα με το να τονίσουμε αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να προαχθούν και να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό αυτούς τους όρους. Και τέταρτον, γενικότερα θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμό και συνέχεια μεταξύ των δύο αυτών προγραμμάτων, ώστε να διασφαλίζεται ότι με μια εναρμονισμένη προσέγγιση ακολουθούνται οι στόχοι ε, των επισητιστικών αναγκών και ακολουθείται ε, ασφαλής ε, επιτυχής διαχείριση. Προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το πρόγραμμα και να τροποποιηθεί με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο εύρος που θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικό τελικά και να παράσχει καλύτερη αξία, μεγαλύτερο όφελος για τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά που χρησιμοποιούνται γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ήταλα, εισηγητής, έχει τον λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από πλευρά μου θα ήθελα να πω ότι είναι απόλυτα σαφή η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για αυτό το θέμα. Και είναι απλό να συναγάγει κανεί τα συμπεράσματά του από αυτή την έκθεση. Τώρα, δεν ασκήθηκε επιρροή, δεν υπήρξε επίπτωση όσον αφορά την εξισορρόπηση της αγοράς δεν υπήρξε κάποια επίτευξη των επισητιστικών στόχων. Αυτές οι επιδοτήσεις για το πρόγραμμα για το γάλα είναι πολύ μικρές. Οι δαπάνες οι γραφειοκρατικές και η επιβάρυνση είναι υπερβολικά μεγάλες ε, προσωπικά ενδιαφέρθηκα όταν στην ίδια μου την πόλη σε μια εφημερίδα διάβασα στο παρελθόν ένα άρθρο και αποφάσισαν μετά οι δημοτικές αρχές της πόλης να καταργήσουν αυτό το πρόγραμμα επειδή είχε πλέον επέλθει ο κόρος για τον διευθυντή του σχολείου αυτού και δεν είχε καθόλου πλέον όρεξη να συνεχίσει υπό τη γραφειοκρατική αυτή επιβάρυνση να αιτείται την επιχορήγηση. Και αλλού στην Ευρώπη το ίδιο συνέβη. Στην πρακτική εφαρμογή υπήρξε η συμπαρέσυρε αυτή η κατάσταση πολλά σχολεία και τώρα όμως γενικά να σταματήσει αυτό το πρόγραμμα συλλήβδιν είναι μια δυνατότητα βέβαια από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να δούμε ότι η αξιοπιστία, το κύρος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα μπορούσε να υποστεί ένα πλήγμα. Από την άλλη πλευρά μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε τα πράγματα, να ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία. Σε εμά τα, τα παιδιά στη Φινλανδία ε, καταναλώνουν αρκετό γάλα. Δεν χρειάζονται επιδοτήσει για κάτι τέτοιο. Σε άλλε χώρε όμω ίσω συμβαίνει κάτι διαφορετικό και πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένη στοχοθέτηση σε συγκεκριμένε περιφέρειε και περιοχέ για να μπορούν τα, οι μαθητέ να καταναλώνουν γάλα. Γιατί κατά τα άλλα θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το πρόγραμμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ, έχει τον λόγο. You presume rightly, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ εσάς, τον κύριο Ιτάλα, τον κύριο Κιούμπικ, όλα τα μέλη αυτής της Επιτροπής για την ευκαιρία που μου δίνετε να ανταλλάξουμε απόψεις για τα προγράμματα του γάλακτος και των φρούτων στα σχολεία, ειδικότερα μετά την ε, δημοσίευση της έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεκτικό συνέδριο, αλλά και τον κύριο Ιτάλα πιο συγκεκριμένα, για τις συστάσεις και τις προτάσεις που έχουν καταθέσει, ώστε τα προγράμματα αυτά να είναι πιο αποτελεσματικά. Εκτιμούμε ιδιαιτέρως τις ε, προτάσεις τους. Το πρόγραμμα για το γάλα στα ευρωπαϊκά σχολεία και το πρόγραμμα για τα φρούτα στα ευρωπαϊκά σχολεία, πέραν του διατροφικού τους χαρακτήρα έχουν και εκπαιδευτικούς στόχους, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να υιοθετήσουν ένα υγιές τρόπο ζωής, να υιοθετήσουν την υγιεινή διατροφή. Ε, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι καλές αυτές συνήθειες τείνουν να μονιμοποιούνται και αργότερα στη ζωή ε, των παιδιών, τα οποία θα γίνουν μετά ενήλικοι. Έχει λοιπόν παιδαγωγική αξία όλο αυτό πέρα της ε, διατροφικής. Προωθώντας την κατανάλωση φρούτων και γαλακτοκομικών προϊόντων, ε, η Επιτροπή επίσης επιθυμεί να υπάρχει μια σωστή ισορροπία ε, στην αγορά ως προς τα προϊόντα αυτά στο πλαίσιο της νομοθετικής πρότασης για την κοινή αγροτική πολιτική, τις μεταρρυθμίσεις δηλαδή που προτείνονται για μετά το 2014 μέχρι και το 2020, η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση του προγράμματος αυτού και προβλέπει αυξημένο προϋπολογισμό της τάξης των 150 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή Είμαστε στα 90 εκατομμύρια ευρώ. Προβλέπεται και η δυνατότητα συγχρηματοδότησης των συνοδών μέτρων τα οποία χρηματοδοτούνται αυτή τη στιγμή πλήρως από τους ε, δικαιούχους. Εμείς προτείνουμε λοιπόν να τα συγχρηματοδοτήσουμε. Η πρόταση αυτή συνάδει με τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Όσον αφορά ε, στο πρόγραμμα για το γάλα στα σχολεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμμερίζεται την αξιολόγηση του ελεκτικού συνεδρίου ως προς το μέγεθος των αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί. Το 2008 και το 2009 έγινε η τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος αυτού μετά από μια μακρά περίοδο διαβούλευσης με τα κράτη-μέλη, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τους λοιπούς αμπλεκόμενους φορείς. Προέκυψαν ε, συστάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, διεύρυνση του καταλόγου των επιλέξιμων προϊόντων, αποκλεισμών αποκλεισμός ορισμένων συστατικών ουσιών κατά την ε, παρασκευή του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι για την υγεία. Έχουν λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα αυτό όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, τα κράτη-μέλη το στηρίζουν. Θα ήθελα να σημειώσω επίσης ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει το πρόγραμμα αυτό από τη στιγμή που συμφώνησε στην αύξηση κατά 9 εκατομμύρια ευρώ ε, των ποσών που ε, επιφυλάσσονται και τίθενται κατά μέρο ε, για το πρόγραμμα αυτό ε, όπως ε, έχει κατατεθεί η πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπής. Δηλαδή από τα 81 εκατομμύρια ευρώ η Επιτροπή πρότεινε να πάει στα 90 εκατομμύρια ευρώ το πρόγραμμα και το Κοινοβούλιο συμφώνησε. Το πρόγραμμα αυτό ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές να συμβάλλουν επιπρόσθετα κεφάλαια έτσι ούτως ώστε να αυξηθεί το τελικό συνόλο της χρηματοδότησης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν ε, την προσχώρηση στο πρόγραμμα αυτό, πολλά κράτη-μέλη δεν είχαν δικό τους εθνικό πρόγραμμα. Λαμβάνοντας τώρα υπόψη τα μέτρα λιτότητας που υιοθετούνται σε διάφορα κράτη-μέλη, η διακοπή του προγράμματος αυτού ουσιαστικά θα σημαίνει την εξαφάνισή του. Και στα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν μέτρα λιτότητας, αλλά και στα υπόλοιπα γενικώ. Ίσως θα έπρεπε ε, να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για να γίνει πιο αποτελεσματικό το πρόγραμμα αυτό του γάλακτος στα σχολεία οι προτάσεις μεταρρύθμισης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την ΚΑΠ πέρα από το 2014 ενσωματώνουν τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και του εισηγητή. Ε, έτσι θα υπάρχει εθνική στρατηγική για την υλοποίηση του προγράμματος και θα μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίζει κριτήρια ε, για την στοχοθέτηση, κάτι το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης. Άλλωστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν και άλλες πτυχές του προγράμματος αυτού που είναι πολύ σημαντικές. Τα, τα προϊόντα που καλύπτονται, παιδαγωγική σκοπή, ε, εκπαιδευτική σκοπή, δικαιούχοι, σχολεία κ.ο.κ. Θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για περαιτέρω συνέργειες μεταξύ των δύο προγραμμάτων, το πρόγραμμα για το γάλα και το πρόγραμμα για τα φρούτα. Η αξιολόγηση των δύο ε, προγραμμάτων, το 12 για το γάλα και το 13 για τα φρούτα, θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία ούτως ώστε να τα βελτιώσουμε διατηρώντας ε, πάντοτε σε λογικό επίπεδο το διοικητικό βάρος ε, που θα πρέπει να φέρουν τα κράτη-μέλη προκειμένου να υλοποιήσουν αυτά τα προγράμματα. Σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, τέσσερα μέλη έχουν ζητήσει ε, το λόγο, πέντε μάλλον. Επειδή έχει περάσει η ώρα, προτείνω δύο λεπτά ε, ο καθένα. Ο κύριο Χατζημαρκάκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω ακούγονται όλα αυτά, το πρόγραμμα είναι πολύ περίπλοκο, λέει, υπερβολικά περίπλοκο και δεν δίνει τα αποτελέσματα που απαιτούνται. Και κάπω βρίσκεται μετέωρο εκκρεμή και ίσω θα έπρεπε λέει να το σταματήσουν. Ένα επιχείρημα έχω εναντίον. Ξέρω ότι υπάρχει απόφαση του 10 που αμφισβητεί ότι η Γενική Διεύθυνση Άγκρη θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά. Τώρα, εκείνο που με ενδιαφέρει είναι η παιδαγωγική πτυχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά η πτυχή τη δημόσια υγεία. Υπάρχουν γι' αυτά εντολή στι συνθήκε Λισαβόνα. Εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε αρμόδιοι για την δημόσια υγεία. Όμω όχι η Γενική Διεύθυνση Άγκρη, αλλά ο κ. Ντάλι για την υγεία των ε, καταναλωτών. Αυτή την πτυχή πρέπει να δούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Μια άλλη πτυχή είναι ο ευδιάκριτος χαρακτήρας τη Ευρωπαϊκής Ένωση, που δεν διασφαλίζεται. Δεν βλέπουν στι καντίνε σχολικέ στα κηλικεία ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Αν θυμηθείτε όμω τι έγινε, τι γινόταν όταν είμαστε μαθητέ, και εγώ το θυμάμαι, υπήρχε σχολικό γάλα, έπρεπε να πληρώνετε. Αν γνώριζα όμω τότε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι που μου δίνει την μπανάνα, όχι την μπανάνα, αλλά το μήλο τέλος πάντων, το φρούτο, τα φρούτα και το γάλα, χωρίς να πληρώνω και μάλιστα σε διαφορά με εκείνα τα οποία αγοράζει κανείς ως μαθητής και που δεν είναι τόσο υγιεινά, τότε αυτό θα ήταν η ιδιαίτερη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα το θυμόμαστε όλοι έτσι. Σε αυτή την περίοδο κρίση είναι πολύ αξιόλογο αυτό το πρόγραμμα για να εγκαταλειφθεί. Πρέπει όμω να μεταρρυθμιστεί εκ βάθρων από ε, τα θεμέλια του. Πρέπει με βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού ε, Δικαστηρίου να αλλάξει η δόμηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτού του προγράμματο και τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τι επιδόσει του. Χωρί δαπάνε, ε, δηλαδή δωρεάν, χωρί επιβάρυνση, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Έτσι να συνεχίσουμε το πρόγραμμα. Θα ήταν πολύ κρίμα να το σταματούσαμε. Απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει απολύτω καινούρια πρόταση. Ευχαριστώ. Mr. Epping, please. κύριος παρακαλώ, έχει τον λόγο. Ναι, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις προς τον κύριο Κούμπεκ. Κούμπικ. Ποιος είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός για τα δύο αυτά προγράμματα, επακριβώς ποια είναι τα νούμερα και δεύτερον, πόσο χρόνο χρειάζε, πόσος χρόνος χρειάζεται ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ενίσχυση τη χρηματική ε, και τελικά να παραδοθεί το γάλα. Πόσος ο χρόνος χρειάζεται για ένα σχόλιο. Ο κύριος Βοτσεχόφσκι παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Από τη μία πλευρά έχουμε φυσικά πλεονάσματα όσον αφορά αυτά τα γεωργικά προϊόντα και έχουν προβλήματα οι γεωργοί να διαθέσουν στην αγορά αυτά τα προϊόντα φρούτα, λαχανικά. Από την άλλη πλευρά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κακές διατροφικές συνήθειες στου αφορά τους πολίτες. Το πρόβλημα έχει διαφορετική εμβέλεια, διαφορετικό εύρος στα κράτη-μέλη. Όμως είναι βέβαιο ότι τα παιδιά σε κάποια σχολεία δεν καταναλώνουν, δεν παίρνουν αρκετά φρούτα. Γι' αυτό το όφελος αυτού του προγράμματος είναι εξόφθαλμο. Και πρέπει να τεθεί το ερώτημα, γιατί δεν λειτουργεί σωστά όπως θα έπρεπε αυτό το πρόγραμμα. Γι' αυτό απευθύνομαι προς το ελεγκτικό συνέδριο. Στρέφομαι στο ελεγκτικό συνέδριο διότι γνωρίζω από την ίδια μου τη χώρα, την Πολωνία, προσωπικά, ότι ίσως υπάρχουν υπερβολικά αυστηρές ε, προδιαγραφές για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος που επιβαρύνουν το πρόγραμμα στην ίδια μας τη χώρα και αυτό καταδείχθηκε και στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Δεν υπάρχει αρκετός αριθμός ε, εμπόρων που να διαθέτουν στα σχολεία αυτά τα προϊόντα και έτσι απέτυχε το πρόγραμμα αυτό. Λοιπόν, παρόμοια προβλήματα υπάρχουν σε άλλα κρατημέλη και αυτό θέλω να το δούμε. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Τι συμβαίνει να δούμε. Δεύτερη μου ερώτηση σε ποιο βαθμό αυτά τα κονδύλια μέσα στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων χρησιμοποιήθηκαν σωστά. Ευχαριστώ. Κυρία Σέσκοβα παρακαλώ. Eh, Σα ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα γενικότερο πλαίσιο, διότι προέρχομαι από μια χώρα όπου ε, κατά την οικοδόμηση του πραγματικού σοσιαλισμού, αυθεντικού σοσιαλισμού, γαλακτοκομικά προϊόντα και τρόφιμα διετίθενται δωρεάν στα σχολεία και το θυμόμαστε αυτό και εγώ το θυμάμαι όταν ήμουν παιδί. Και πρέπει να πω ότι από το, τα δικά μου βιώματα οι επιπτώσεις ε, οι ε, πρέπει να δούμε ότι είναι αρκετά θα έλεγα αποδυναμωμένες ή αμφισβητήσιμες. Θα έπρεπε τα, οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών στα χέρια των γονιών τους και στις οικογένειές τους να βρίσκονται και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζω λοιπόν εγώ την έκθεση, χαιρετίζω την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υποστηρίζω και εστερνίζω με τα συμπεράσματα του εισηγητού από πλευρά του εγγράφου του που κάνουν λόγο για την δυνατότητα κατάργησης πλέον αυτού του προγράμματος συνολικά. Συλλήβδην κατάργηση, όχι δηλαδή μεταρρύθμιση ή ε, νέα προσπάθεια. Επίσης όσον γίνεται, ε, καθώς γίνεται λόγος για διασπάθηση κονδυλίων των φορολογουμένων υποστηρίζω ιδιαίτερα έντονα αυτή τη ε, δράση να καταργηθεί αυτό το πρόγραμμα. Το να υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσει δημοσιονομικά από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών υπό τη σημερινή συγκυρία κρίσης είναι απόλυτα περιττό. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Χολμάιερ παρακαλώ. Εγώ Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να θέσω το ερώτημα μετά από την ομολογία του ΔΕΚ. Σωστά, με πληροφόρησαν σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΚ δεν είναι πλέον δυνατό όταν δεν έχουμε πλεονασματικές παραγωγές, κάτι το οποίο δεν είναι πλεονασματικό, παρόλα αυτά να το διαθέτουμε σε ένα κοινωνικό πρόγραμμα και να πληρώνεται από τον προϋπολογισμό της Γεωργίας, ε, από τα κονδύλια για τη Γεωργία. Καθότι γνωρίζω δεν είναι δυνατό να γίνεται αυτό. Κοινωνικά προγράμματα να πληρώνονται, να καλύπτονται στις ανάγκες τους από τον προϋπολογισμό για τη Γεωργία. Αν δεν υπάρχει κιόλα και πλεονασματική παραγωγή όσον αφορά την διάθεση αυτών των πλεονασματικών προϊόντων στην αγορά, για παράδειγμα σε σχέση με το γάλα για τα παιδιά, για τους πιο φτωχούς να διανέμεται στα σχολεία π.χ. υπό αυτό το πλαίσιο. Δεύτερον, θα ήθελα να θέσω το ερώτημα για τον αριθμό σχολείων και παιδιών που καταφέραμε να προσεγγίσουμε. Δεν μπορούσα να δω ποια είναι, ποιο είναι το εύρος αυτού του προγράμματος. Τρίτον, όταν θέλει κανείς να τολμήσει να κάνει ένα τέτοιο πρόγραμμα πρέπει να διαρωτηθεί είναι σκόπιμο σε σχέση με την υλοποίησή του στο τέλος τέλος τα κράτη-μέλη να μην υλοποιούν όλες αυτές τις διατάξεις. Το είδα στη δική μου χώρα. Την επιμελητιακή υποστήριξη πρέπει να την πληρώνουμε εμείς. Δηλαδή το παιδί πληρώνει για το μήλο ή το αχλάδι που του δίνουμε. Στο τέλος τέλος στη σύγκριση δηλαδή με, την, με το στόχο είναι πολύ μικρά τα αποτελέσματα. Πενιχρά. Κοστίζει εξίσου ένα μήλο σε σχέση με το, εκείνο που αγοράζει κανείς. Γι' αυτό το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ συρρυκνωμένο, πολύ μειωμένο. Στη χώρα μου δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερη επίπτωση αυτό και γι' αυτό σταματήσαμε με αυτό το πρόγραμμα. Επειδή οι ενώσεις λιανικού εμπορίου έχουν καλύτερη μελητιακή υποστήριξη και στο τέλος έχουν πιο προσιτές τιμές για την διάθεση τέτοιων προϊόντων από ότι εμείς που με την κοινωνική μας, ας το πω έτσι, ε, με τα κοινωνικά μας ιδανικά θέλαμε να αλλάξουμε τις διατροφικές συνήθειες των των παιδιών και να τα υποστηρίξουμε να τρώνε φρούτα κτλ. Έχω αμφιβολίε και αν αυτό είναι έργο τη ευρωπαϊκή Επιτροπή και με ποια ανάλυση καταλήγουμε στο να διανέμουμε τέτοια προϊόντα. Είναι αμφισβητήσιμο όμω αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και νομικά δεν μπορεί να ευσταθήσει. Γκάιερ παρακαλώ. Ναι, και από την ίδια χώρα προέρχομαι, όπω έχει η κυρία Χολμάια, όμω από άλλο κρατήδιο, ομοσπονδό κρατήδιο. Στη Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία, λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα. Δεν πληρώνουν τα παιδιά εκεί για τα μήλα και τα χλάδια. Φαίνεται να οφείλεται για το ότι η ελεύθερη, το ελεύθερο κρατήδιο ε, της Βαβαρίας διοργανώνει αυτή την προσπάθεια με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στη Βορεια Ρινανία Βεσφαλία. Εμείς μπορέσαμε να έχουμε σχολεία που ε, μπορέσαμε να προσελκύσουμε να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα για τα κριτήρια ποια σχολεία θα υποστηρίζονται και θα υποστηριχθούν και ήταν από πλευράς ε, της ε, ε, περιφερειακής κυβέρνησης του κρατηδίου αυτή η απόφαση που ελήφθη. Οφείλεται στο ότι έχουμε το τα κοινωνικά έσοδα και το ότι αν αυτά τα προγράμματα όταν διατίθενται δωρεάν έχουν προτέρημα διατροφικό σε σχέση με τα, τους γονείς τους που θα τους στέλνανε ε, με δύο ευρώ στο σχολείο για να αγοράσουν στο τέλος τέλος κάποια σοκολάτα από το κηλικείο. Λοιπόν, μπορούμε να συζητήσουμε αν ως θέμα ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει κάτι τέτοιο ή όχι. Να συμμετάσχω και εγώ σε αυτή τη συζήτηση ευχαρίστω. Αλλά όταν καταλήγουμε στην απόφαση για την κατανομή τέτοιων προγραμμάτων, αν θυμάμαι καλά τον όγκο, 180 εκατομμυρίων ευρώ δηλαδή 90 εκατομμύρια για το ένα και το άλλο πρόγραμμα, να τα σταματήσουμε και να τα σταματήσουμε επειδή τι θα γίνει, θα απελευθερωθούν μικρότερα κονδύλια δηλαδή. Τώρα αν με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετείται συνολικά η γεωργία πανευρωπαϊκά, τουλάχιστον όσον αφορά τον, χρηματοοικονομικό όγκο των φρούτων, δεν είναι κάτι το θετικό μια και υποφελούνται τα παιδιά και γι' αυτό είμαι υπέρ αυτού που είπε ο Γιώργος Χαζημαρκάκης πιο πριν. Μια παρατήρηση στο περιθώριο πρόεδρε αν μου επιτρέπετε. Η, η Ελεύθερη Βαβαρία έχει ήδη δωρεάν γεύμα για όλους. Γι' αυτό είναι θα έλεγα περιτό αυτό το πρόγραμμα για ένα ε, τέτοιο πρόγραμμα φρούτων. Εσείς παρακαλώ έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα εδώ να πω ότι υπάρχουν σίγουρα διαφορετικές εμπειρίες στα διαφορετικά κράτη. Στη Δανία θέλω εγώ να πω ότι υπήρξαν επικρίσεις όσον αφορά το πρόγραμμα φρούτων, διανομής φρούτων στους μαθητές στα σχολεία. Διότι υποστηρίζονται έτσι τα οικονομικά ισχυρότερα σχολεία τα οποία βρίσκονται στις καλύτερες συνοικίες και είναι προνομιούχοι οι μαθητές σε αυτά τα σχολεία. για φρούτα τα οποία διανέμονται, ε, φρούτα που ε, πηγαίνουν σε αυτά τα σχολεία προνομιούχων μαθητών δεν παίρνουν τα φρούτα άλλα σχολεία όπου είναι οι μαθητές με τις περισσότερες ανάγκες αποκλείονται αυτοί οι μαθητές ε, μέσα από αυτές τις διαδικασίες και ασκήθηκε, ασκήθηκαν επικρίσεις για αυτή την κατάσταση στη Ιδανία. δεν είναι ιδιαίτερα θετικά λοιπόν τα πράγματα Υπάρχουν ίσως κάποιες δυνατότητες για την υγιεινή διατροφή των παιδιών και έτσι πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, διαφορετικές απόψεις ακούστηκαν. Πρώτα θα δώσω τον λόγο πάλι στο ελεγκτικό συνέδριο να απαντήσει τα ερωτήματα και να σχολιάσει στις παρατηρήσεις που έγιναν. Κύριε Κούμπικ, έχετε τον λόγο παρακαλώ. I will start... Ε, Μάλιστα, ευχαριστώ και θα ξεκινήσω με κάποιες γενικές παρατηρήσεις πρώτα που αφορούν τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος για το γάλα ε, εξειδικευμένα και τι θα πρέπει να κάνουμε με αυτό το πρόγραμμα. Θέλω να τονίσω, να υπογραμμίσω εδώ κάτι. Αυτό που εκφράσαμε εμείς στην έκθεσή μας δηλαδή. Ιδιαίτερα με τη σημερινή μορφή του προγράμματος για το γάλα στα σχολεία που πολύ λίγα επιτυγχάνει, πολύ πενιχρά τα αποτελέσματα. Η επιβάρυνση γραφειοκρατική σε σχέση με τις δαπάνες είναι υπερβολική και δεν έχουμε κανένα θετικό όφελος όσον αφορά την κατανάλωση γάλακτος από τα παιδιά του μαθητέ στα σχολεία. Η καλύτερη εναλλακτική λύση για το γάλα είναι να υπάρξει σε βάθος εκθεμελίων μεταρρύθμιση ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει μέσα σε ένα νέο πλαίσιο η άποψη, αν αυτή αν υιοθετηθεί, αν υπάρξει αυτή η προοπτική, τότε θα μπορούσε να διατηρηθεί αυτό το πρόγραμμα. Πρόκειται για την απόφαση από τα αρμόδια όργανα που θα έπρεπε να λάβει αυτή την κατάσταση πραγμάτων υπόψη. Μπορώ να πω ότι έκανε σωστά τη δουλειά το ελεγκτικό συνέδριο, διατύπωσε συστάσεις που εφ' τώρα είναι δημόσιες, έχουν δημοσιοποιηθεί και μπορούν να είναι στη διάθεση των Ευρωβουλευτών για να εξεταστούν. Τώρα για τον προϋπολογισμό θα ήθελα να πω κάτι. Το σημερινό επίπεδο δαπανών όσον αφορά το 2011 είναι περίπου 180 εκατομμυρίων ευρώ η κατάσταση των δύο προγραμμάτων δεν είναι ακριβώ η ίδια κατά το ίμιση το ένα και κατά το ίμιση το άλλο. Το ένα πρόγραμμα λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια όπω είπα και έχει ένα σταθερό επίπεδο δαπανών περίπου 70 εκατομμυρίων. Ε, το άλλο πρόγραμμα για τα φρούτα είναι στην πρώτη του φάση. Ε, το, τα 90 εκατομμύρια δεν χρησιμοποιήθηκαν πλήρως το 2010 λόγω της καθυστερημένης έναρξης αυτού του προγράμματος. Όμως ε, αυτή η δαπάνη θα αυξηθεί, το κονδύλιο αυτό θα αυξηθεί. Για κάποια τώρα αυστηρά πλαίσια εθνικών κανόνων και κανονισμών θα, λάβει τον λόγο, θα λάβουν τον λόγο να τοποθετηθούν οι συνάδελφοί μου ελεγκτέ του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα ήθελα να τονίσω όμω για άλλη μια φορά ότι το κύριο συμπέρασμά μα και το κύριο μήνυμά μα είναι να βελτιωθούν αυτά τα προγράμματα. Όχι να καταργηθούν, αλλά να βελτιωθούν. Και έχουμε πολύ καλά παραδείγματα με βάση την αξιολόγηση του προγράμματο για τα φρούτα. Το πρόγραμμα για τα φρούτα είναι μια καλή εμπειρία. Έχουμε θετική πείρα και για την επιλογή για τις βελτιώσεις που μπορούν να επιτευχθούν προς την ίδια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί και το πρόγραμμα για το γάλα στα σχολεία. Μάλιστα, θα ήθελα να πάρουν το λόγο οι συνάδελφοί μου για να σας δώσουν κάποιες ε, πιο εξειδικευμένες ε, πληροφορίες σε θέματα ε, λεπτομεριακά. Θα ήθελα να τονίσω γενικά ότι αληθεύει ότι η πείρα μας σε σχέση με τις χώρες τα βιώματα που έχουμε είναι πολύ διαφορετικά από χώρα σε χώρα και στην έκθεσή μας μπορείτε να βρείτε σίγουρα κάποια πολύ καλά παραδείγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης και σε σχέση με άλλες χώρες ως θετικά παραδείγματα. Κάνουμε λόγο τώρα για την Πολωνία. Η Πολωνία είναι ένα παράδειγμα μιας χώρας που έκανε χρήση κάποιων πρακτικών που μπορούν να θεωρηθούν καλές πρακτικές σας ευχαριστώ. Ο Διευθυντής κύριος Προμιάσκη, παρακαλώ. Ε, το εκτιμώ ότι θέλει να επιθυμήσει, το, να απαντήσει το δυνατόν λεπτομερέστερα αυτά τα θέματα το ελεγκτικό συνέδριο, μόνο που πίεζε ο χρόνος. Παρακαλώ να είσαστε συντομότατος. Ευχαριστώ. Ναι, Πρόεδρε, θα είμαι και το υπόσχομαι συντομότατο. Για τα ερωτήματα, τι ερωτήσει που έγιναν για τον ετήσιο προπολογισμό, ήταν 74 εκατομμύρια για το γάλα και 90 εκατομμύρια για τα φρούτα πολύ λιγότερα δαπανήθηκαν για τα φρούτα. Επειδή είχαμε προβλήματα στην πρώτη αυτή φάση υλοποίηση του προγράμματο για τα φρούτα και στην ερώτηση του κυρίου Βοτσεχόφσκι, αν είναι δυνατόν να βρεθούν περισσότερε λεπτομέρειε για τι σημερινέ δαπάνε, ναι. Είναι, έχουμε το παράρτημα 4 στην έκθεση, όπου ενδεικτικά αναφέρουμε τι δαπανήθηκαν ανά κράτος μέλος. Αν έχετε ανάγκη για πιο εξειδικευμένα στοιχεία, είμαστε στη διάθεσή σα να τα παράσχουμε. επίση και η Επιτροπή μπορεί να το κάνει. Για το άλλο εξειδικευμένο ερώτημα, πόσο χρονικό διάστημα παίρνει η επεξεργασία ενός φακέλου του γραφειοκρατικού βάρους δηλαδή. Εδώ πρέπει να πούμε δεν υπάρχει μία ενιαία και μόνη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Εξαρτάται από το πρότυπο διανομής που υιοθετείται από ένα κράτος μέλος. Εξαρτάται από το κράτος μέλος. Πώς δηλαδή συμπληρώνονται αυτές οι αιτήσει ε, δύο φορές ε, ανά έτος σχετικά απλό. Και ακόμα και αυτή η απλή υποχρέωση είναι υπερβολική επιβάρυνση για τα σχολεία σε σχέση με τα κονδύλια που διατίθενται. Οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των σχολείων λένε δεν θέλουμε να τα συμπληρώνουμε όλα αυτά γιατί παίρνουμε 50 ή 100 ευρώ σε επιστροφή. Σε άλλες ε, ε, χώρες είναι πολύ πιο δαπανηρές ε, από πλευρά χρόνου αυτές οι διεργασίες. Εξαρτάται από τα κράτη-μέλη πώς διοργανώνουν αυτά τα πλαίσια, τα γραφειοκρατικά ε, τώρα για το πόσα σχολεία και πόσοι μαθητές επωφελήθηκαν από αυτά τα προγράμματα όπως ρωτήθηκε για το γάλα ενδεικτικά 10% είναι η πιθανή, ε, ο πιθανός αριθμός των μαθητών που επωφελήθηκε δυνάμει από αυτό το πρόγραμμα Στατιστικά ίσως δεν αντανακλάται απόλυτα η πραγματικότητα, αλλά δεν έχουμε άλλα στοιχεία για το, τα φρούτα δεν ήταν δυνατό σε αυτή τη φάση σύνταξη τη έκθεση να πούμε πόσοι μαθητέ επωφελήθηκαν, γιατί μόλι είχε ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό για τα φρούτα. Για την επιμελητιακή υποστήριξη και το κόστο δαπάνη επιμελητιακή υποστήριξη υπάρχει κάποια επιβάρυνση που και αυτήν όμω ε, αναλαμβάνουν τα εθνικά, ε, οι εθνικές δημοσιονομικές αρχές. Αυτό που έχει αξία είναι να διανέμονται τα φρούτα στους ε, εκείνους που έχουν ανάγκη και πρέπει να υποφεληθούν τους μαθητές σε σχέση με τις ε, τιμές ε, που, στις οποίες ήταν διαθέσιμα αυτά τα προϊόντα όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Βοητσεχόφσκι για τους ε, αυστηρούς κανόνες ε, που υιοθετούνται από τις πολωνικές αρχές και πάλι εδώ τα κράτη-μέλη είχαν την ελευθερία διακριτικής ευχέρειας ε, να επιλέξουν το τι θα έκαναν. Βλέπουμε εδώ ένα παράδειγμα ανάγλυφης γραφειοκρατικής επιβάρυνσης σε σχέση με τις τους Σε άλλα κράτη-μέλη κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβαίνει το επίπεδο επιβάρυνσης είναι αρκετά υψηλό σε όλα τα κράτη-μέλη. Και αυτό ως ε, ε, ε, εν μέρη απάντηση, γιατί το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε με καθυστέρηση, όπως προανέφερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σκούμπικ. Για να ολοκληρώσω, Πρόεδρε, επειδή αρχικά ήταν έγιναν σχόλια από δύο άτομα όσον αφορά την στοχοθέτηση, τη στοχοθετημένη ομάδα. Είναι αναγκαία η στοχοθέτηση για να έχει αποτελέσματα αυτό το πρόγραμμα, αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συγκυρία τουλάχιστον. Ένα μέρος πηγαίνει εκεί όπου δεν είναι τόσο χρήσιμο ή εκεί όπου δεν το χρειάζονται ιδιαίτερα. Και αυτό το παρουσιάσαμε ως παρατήρηση στην σελίδα 22 στην έκθεσή μας αν θέλετε να στοχοθετήσετε, θα πρέπει να στοχοθετήσετε ε, με αποτελεσματικό τρόπο, με εξειδικευμένο τρόπο. Ο πιο εξειδικευμένος τρόπος στοχοθέτησης είναι ο πιο δαπανηρός. Πρέπει να βρούμε όμως ε, μια σωστή ισορροπία μεταξύ του κόστους επιβάρησης και τη στοχοθέτηση και τα αποτελέσματα που μπορούμε να πετύχουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στοχοθέτηση, πράγμα το οποίο ίσως μπορεί να φαίνεται φθηνότερο, αλλά είναι όμως πολύ χαμηλής επίδοσης, με πολύ χρέση επιδόσει και αυτό πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Η Επιτροπή πολύ σύντομα, παρακαλώ. Yes, Mr. Chairman, I will be very brief. είμαι πολύ σύντομο, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ε, ελέγχθη κάτι για την όλη ορατά του προγράμματων. Στα διάφορα προγράμματα επιστημικά είναι υποχρεωτικό να γνωρίζουμε από πού προέρχονται τα χρήματα που αφορά τα παιδιά. Ποιο κάνει δηλαδή την επιδότηση. Και για το γάλα πρέπει να υπάρχει ένα πόστερ και να εξηγούνται τα πάντα στα σχολεία. Τώρα, αν το βλέπουν τα παιδιά να το προσέχουν, είναι άλλο θέμα. Επίσης, απαντήθηκαν διαφορά, πρέπει να σα πω ότι το 2010 δόθηκαν 70 εκατομμύρια και για τα φρούτα 53 εκατομμύρια Έχουμε λοιπόν σε σχέση με τα προβλεπόμενα εκατομμύρια λιγότερα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, ιδιαίτερα για το πρόγραμμα που αφορά τα φρούτα. Επίσης τέθηκε ένα θέμα για τους πολύπλοκους κανόνες, απήντησε το ελεγκτικό συνέδριο και εγώ μπορώ να επιβεβαιώσω ότι όντως ε, είναι στη εκκριτική ευχαίρεια των κρατών μερών να εκτελέσουν το πρόγραμμα αυτό σύμφωνα με τους κανόνες τους και πολλές φορές όντως τα πράγματα είναι κάπως πολύπλοκα. Επίσης, μια άλλη ερώτηση ήταν σε ποιο μέτρο θα πρέπει τα σχολεία να εκπαιδεύουν τα παιδιά για την υγιεινό τρόπο διατροφής και ζωής, ιδιαίτερα για τα φρούτα. Έχουμε συνοδευτικά μέτρα με τα οποία προσπαθούμε να εμπλέξουμε στο μέτρο του δυνατού στο όλο πρόγραμμα και τους γονείς. Δηλαδή, εκπαιδεύονται τα παιδιά να φέρουν και φρούτα από το σπίτι τους. Και έτσι ασκούν πίεση στους γονείς για να συμμορφωθούν με τη γενικότερη ε, συνήθεια που επικρατεί στο σχολείο. Μετέχουν λοιπόν και οι γονείς. Όσον αφορά το θέμα της νομικής βάσης, είναι πρόγραμμα που αφορά τους ε, λιγότερο, τους περισσότερο ενδεείς και δεν νομίζω ότι εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για διακριτική ευχαίρεια του κάθε κρατήματο. Τόσο αφορά τον αριθμό των παιδιών, σύμφωνα με του δικού μα αριθμού, για τα φρούτα στο σχολείο. Μιλάμε για 5 εκατομμύρια παιδιά και για το γάλα, παρά το γεγονό ότι αφορά το 10% του πληθυσμού, έχουμε να κάνουμε με 21 εκατομμύρια παιδιά. Δεν είναι αμελητέ αυτέ οι ποσότητε. Όσον αφορά τώρα το θέμα τη επιμελητία και ποιο πληρώνει, την προσφορά που γίνεται για να δοθούν τα φρούτα και το γάλα στο σχολείο, συμπεριλαμβάνεται αυτό το κόστος. Το κόστος μεταφοράς μπορεί να είναι maximum το 3% του κόστους του ολικού για την ε, παροχή των φρούτων. Τώρα, στόχευση. Τελευταία ερώτηση. Όπως είπα ήδη στην εισαγωγική μου παρατήρηση, υποβάλαμε πρώτα στο Συμβούλιο ώστε και το θέμα αυτό να συζητηθεί ώστε να υπάρχει καλύτερη στόχευση. Δηλαδή τα σχολεία τα οποία έχουν περισσότερο ανάγκη από τέτοιου είδους μέτρα. Κύριε Ήταλα, θέλετε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με εσάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, το πρόγραμμα αυτό για τα φρούτα είναι σωστά στοχευμένο και δουλεύει σωστά. Το πρόβλημα είναι με το πρόγραμμα για το γάλα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι, ότι με διαφορετικούς στόχους. Ο πρώτος είναι να δούμε πώς δουλεύει ο γαλακτοκομικός τομέας και αγορά και εδώ υπάρχουν ε, προβλήματα. Και νομίζω ότι έτσι όπως ε, γίνεται το πρόγραμμα δεν υλοποιούμε τους στόχους μας διότι έχει γενικότερα. Πιστεύω ότι πρέπει καλύτερα να στοχεύσουμε και κυρίως να δούμε σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ποιες είναι οι ανάγκες για να έχουμε καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση του θέματος αυτού. Περνούμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης ε, πώς βλέπουμε τις εξελίξεις ε, στο θέμα της ε, οργάνωσης και διαχείρισης στην ε, χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερως στα πλαίσια της άσκησης απλοποίησης του όλου συστήματος. Είστε δύο, έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Πέντε λεπτά ο καθένας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η μελέτη για τα μέτρα πλούστευσης των διαρθρωτικών ταμείων, την οποία διενεργήσαμε τους τελευταίους τρεις μήνες, κατέληξε σε συγκεκριμένες ε, ε, μεθόδους και σε συγκεκριμένους στόχους, στους οποίους θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία και στη συνέχεια θα προβάλλω τα συμπεράσματα και τις συστάσεις. Ε, αναλύσαμε πολύ το θέμα των δικαιούχων. Στο παρελθόν είχαμε αναλύσει το σύνολο των κανόνων, ε, το πώς διαχειρίζονται την κατάσταση οι ελεκτικές αρχές. Ε, μας ενδιαφέρει και η άποψη των δικαιούχων. Η μελέτη διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια τριών μηνών και έτσι δεν μπορέσαμε να εξετάσουμε όλους τους τροποποιητικούς κανονισμούς που εισήγαγαν μέτρα απλούστευσης. Γι' αυτό και μας ενδιέφερε βασικά το εξής. Οι τρεις επιλογές απλουστευμένου ε, κόστους, αν θέλετε, για να βελτιώσουμε την κατάσταση για τους δικαιούχους, προκειμένου να τους καταβληθούν οι δαπάνες χωρίς να πρέπει να ε, υποβάλουν επαχθές υλικό τεκμηρίωσης. Μας ενδιέφερε επίσης ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα μέτρα απλούστευσης στον τομέα της έρευνας και των τεχνολογικών εξελίξεων. Κάναμε πολλές διαβουλεύσεις στα κράτη-μέλη, Αυστρία, Βέλγιο, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο. Με όλες αυτές τις χώρες είχαμε διαβούλευση, μιλήσαμε με τους δικαιούχους, με τις διαχειριστικές αρχές και στη συνέχεια ζητήσαμε τη Συμβουλή της Γενικής Διεύθυνσης για τις Περιφέρειες αλλά και της Γενικής Διεύθυνσης για την Απασχόληση. Ποια είναι τα βιώματα των Γενικών Διευθύνσεων, ποιες είναι οι εμπειρίες και οι προσδοκίες τους. Και στο τέλος κάναμε μια έρευνα στην οποία συμμετείχαν 87 διαχειριστικές αρχές από 23 κράτη-μέλη ε, και έτσι μπορέσαμε να συλλέξουμε τις απόψεις τους. Μια πρώτη εικόνα του πώς λειτουργούν όλα αυτά είναι αυτή που βλέπετε στην οθόνη. Εδώ βλέπετε το βαθμό στον οποίο τα μέτρα απλούστευσης, αυτές οι τρεις, τρεις απλουστευμένες επιλογές κόστους, ουσιαστικά μεταφράστηκαν και ενσωματώθηκαν στην Εθνική Νομοθεσία για την Επιλεξιμότητα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε αυτό το εξής. Αν υιοθετήσει η Επιτροπή ένα κανονισμό για τους κανόνες επιλεξιμότητας, αυτοί ε, δεν είναι διαθέσιμοι οι κανόνες άμεσα για τους δικαιούχους. Πρέπει ε, να το ενσωματώσει αυτό το κράτος μέλος τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας πριν μπορέσει ο εκάστοτε δικαιούχος να αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο. Πιστεύουμε σε γενικές γραμμές ότι τα μέτρα πλούστευσης έχουν πολύ μεγάλο δυναμικό δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό αυτό ακόμα. Με μπλε βλέπετε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με πράσινο βλέπετε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Βλέπετε πολλές διαφορές ε, ως προς το πόσο έχουν ε, ακολουθηθεί αυτές οι επιλογές ε, απλούστευσης. Η Αυστρία είναι ενθουσιώδης οπαδός της απλούστευσης, για παράδειγμα, ενώ προχωρώντας προς τα δεξιά από τη μεριά του γραφήματος βλέπουμε ότι άλλα κράτη-μέλη έχουν επιλέξει πολύ λιγότερο την απλουστευμένη άγουσα, την απλουστευμένη αυτή οδό για το ΕΚΤΑ και το ΕΤΠΑ και έξι κράτη-μέλη δεν έχουν καν υιοθετήσει αυτή την επιλογή την απλουστευμένη. Ε, και μάλιστα χώρες που αξιοποιούν ιδιαίτερο στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή το ΕΤΠΑ, όπως η Ισπανία και η Πολωνία. Σε γενικές γραμμές εκτιμούμε ότι το 55% του συνόλου των πόρων του ΕΚΤΑ καλύπτονται και το 8% του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ. Επομένως, προκειμένου να είναι πιο σαφής η διαδικασία με την οποία ενσωματώνονται αυτές οι επιλογές στην εθνική νομοθεσία, ο συνάδελφος θα μας μιλήσει για την αυστριακή εμπειρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Αυστρία ήταν μία από τις πρώτες χώρες που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Ουσιαστικά λειτουργήσε ως πρωτοπόρος τρόπον την Α. Αν δείτε αυτή την, αυτό το πίνακα, βλέπετε τι έχει γίνει από το Μάιο του 2009 μέχρι τον Οκτώβριο του 2010. Χρειάστηκε η Αυστρία 1,5 χρόνο για να ενσωματώσει, να εφαρμόσει αυτό τον ευρωπαϊκό κανονισμό και να τον... Ε, μετατρέψει σε μια ε, τρέχουσα εθνική πρακτική Εάν δείτε τις μελέτες που, ε, τις μελέτες που έχουν γίνει για το θέμα αυτό, το συμπέρασμα είναι ότι η διαδικασία απλούστευσης χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο και δεν ήταν και καθόλου εύκολη. Η απλούστευση δηλαδή δεν ήταν καθόλου απλή. Χρειάστηκε ένας χρόνος να συνταχθεί πρόταση, πόσο μάλλον να καταλήξουμε σε οριστική εκδοχή. Οι αυστριακές αρχές θεωρούν ότι η διαδικασία απλούστευσης ε, προσθέτει στο διοικητικό άχθος, κυρίως λόγω κάποιων αβεβαιοτήτων οι οποίες παραμένουν. Βλέπετε ότι στις 15 ε, Οκτωβρίου του 2010 ε, οργανώθηκε αυτό το εργαστήριο διάδοσης ε, και δημοσιοποίησης αυτής της επιλογής της απλουστευμένης Υπήρχαν δηλαδή ακόμα αμφιβολίες για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν όλες αυτές οι διατάξεις. Ο προηγούμενος ομιλητής παίρνει τη σκητάλη και λέει «Να σας δώσω κάποιες λεπτομέρειες για αυτά τα ε, μέτρα γενικότερα». Ε, οι διαχειριστικές αρχές μας έχουν ε, εκφράσει όχι τόσο μεγάλο θεσουριασμό όσο θα περιμέναμε. Δεν έχουν υπάρξει αλλαγές με αυτά τα μέτρα απλούστευσης δεν έχει μειωθεί το διοικητικό άχθος των διαχειριστικών αρχών ούτε των δικαιούχων. Ένα τέταρτο των απαντώντων θεωρεί ότι η διαδικασία όντως είναι πολύ πιο εύκολη, ενώ άλλοι θεωρούν ότι ενδεχομένω ε, η διαδικασία έχει γίνει πιο περίπλοκη. Τώρα, ε, αυτό για τα μέτρα απλούστευσης. Ως προς τις επιλογές απλουστευμένου κόστους, η κατάσταση είναι πολύ πιο θετική. Ε, πολύ περισσότεροι θεωρούν ότι έχει μειώσει το διοικητικό άχθος. Από το 50% μέχρι το 70% όσων απάντησαν θεωρούν αυτοί ότι όντως συμβάλλει στη μείωση ε, του διοικητικού φόρτου. Ε, και για τους δικαιούχους ισχύει αυτό και για τις διαχειριστικές αρχές. Το 67% των δικαιούχων θεωρεί ότι όντως μειώνεται το διοικητικό ε, φορτίο και πολύ μικρό προσωστό αυτών που απάντησαν θεωρούν ότι αυξάνεται το διοικητικό ε, βάρος. Και βεβαίως αρκετοί δεν γνωρίζουν ακόμα ε, τι συνεπάγεται όλη ε, αυτή η καινούργια επιλογή, η πιο απλουστευμένη. Είναι λογικό αυτό, γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει ούτε είναι απολύτως γνωστό σε όλους. Θα γίνει πιο αποτελεσματική αυτή η επιλογή στο μέλλον. Ε, ένα σαφές όφελος τόσο για τις διαχειριστικές αρχές όσο και για τους δικαιούχους είναι η λιγότερη ε, χαρτούρα αν θέλετε. Δηλαδή περισσότερος χρόνος αφιερώνεται στην υλοποίηση της διαδικασίας και πολύ λιγότερο στη συμπλήρωση διαφόρων εντύπων και υποβολή. Ε, το θέμα είναι αν επηρεάζονται τα ποσοστά συμμετοχής. Οργανώσεις που πίστευαν στην, στο παρελθόν ότι είναι πολύ πολύπλοκη διαδικασία και δεν συμμετείχαν, τώρα συμμετέχουν περισσότερο. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι μικρές οργανώσεις, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι μικρές οντότητες γενικότερα τώρα συμμετέχουν πιο ενεργά ε, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε πολύ θετική ανατροφοδότηση, πολύ θετικό feedback από τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις τα ερευνητικά ιδρύματα και οι οργανισμοί τοπική αυτοδιοίκησης δεν έχουν επωφεληθεί τόσο από, αυτά, από αυτές τις επιλογές απλούστευσης. Για τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα ο λόγος βασικά είναι τα κατόφλια, τα οποία είναι πολύ χαμηλά. Αυτό θέλουμε να τονίσουμε. Αυτό έχει να κάνει με το σχεδιασμό των μέτρων εξ αρχής. Θεωρούνται τα κατόφλια χαμηλά γενικότερα για την, ε, την αποκοπή, την εφάπαξη καταβολή του ποσού, το όριο είναι το 20%. Πολλοί από όσους απάντησαν και πολλοί από τους συνεντευξιαζόμενους ε, που προέρχονται από την έρευνα και από τα πανεπιστήμια επισημαίνουν ότι συνήθως τα κόστη είναι πολύ υψηλότερα από αυτό το ποσοστό. Επίσης κάποιες παρατηρήσεις έχουν γίνει ως προς τη διαδικασία. Οι διαχειριστικές αρχές μας λένε ότι ε, έχοντας φτάσει στα μέσα τους προγράμματος, ε, υπησέρχονται τα μέτρα απλούστευσης. Καλά είναι, αλλά εμείς έχουμε συντάξει ήδη όλα τα εγχειρίδια και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσουμε το εγχείρημα από την αρχή, ε, αναφέροντας το πρόγραμμα, διαδίδοντας όλα αυτά τα νέα και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό λοιπόν πολλές διαχειριστικές αρχές δεν έχουν αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία, γιατί ήδη βρίσκονται στα μισά του δρόμου. Και ε, οι μεθοδολογικές απαιτήσεις είναι κάποιος περίπλοκες και αυτό συνεπάγεται καθυστερήσεις και έλλειψη ενδεχομένως νομικής ε, βεβαιότητας. Ε, για το αν μπορεί κανείς να υποβάλει αιτήσει πρώτης πληρωμής χρησιμοποιώντας αυτή την απλουστευμένη επιλογή. Τώρα, ως προς το θέμα της Αυστρίας, παρά το γεγονός ότι η Αυστρία λειτουργήσε πρωτοποριακά και ήταν η πρώτη ίσως χώρα που ε, ε, εφήρμοσε ε, αυτή τη διαδικασία, η εμπειρία μας είναι ακόμα περιορισμένη. Δεν είναι επαρικής ίσως. Άλλωστε, οι επιλογές αυτές δεν έχουν ακολουθηθεί από αρκετά μεγάλο ποσοστό των τελικών αποδεκτών. Δεν είναι δηλαδή ε, αρκετά γνωστό και έτσι δεν έχουμε αρκετά στοιχεία πάνω στα οποία να μπορούμε να βασιστούμε. Δεν το γνωρίζουν αυτό παρκώς οι δικαιούχοι, ποιες είναι οι ευκαιρίες δηλαδή που τους προσφέρονται με αυτές τις διαδικασίες της απλούστευσης. Ενδεχομένως υπάρχει μια κάποια διαφορά μεταξύ διαχειριστικών αρχών και δικαιούχων. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε για την Αυστρία είναι ότι έχουμε ε, μια σχετική μείωση του βάρους, όχι πολύ μεγάλη και για τις διαχειριστικές αρχές. Σίγουρα εξοικονομούν στο στάδιο των πληρωμών, ωστόσο αυτό αντισταθμίζεται, αν θέλετε, από αυξημένο βάρος στο στάδιο των αιτήσεων Πάρα πολλά πράγματα πρέπει να επαληθευτούν και να ελεγχθούν από τη διαχειριστική αρχή κατά το στάδιο της υποβολής της αίτηση. Όντως πληρούν με τις προϋποθέσεις οι δικαιούχοι αυτοί, ε, ούτως ώστε να ακολουθηθεί η απλουστευμένη διαδικασία. Οι ίδιοι δικαιούχοι από την άλλη θεωρούν ότι τα κατόφλια είναι εξαιρετικά χαμηλά για να καλύψουν τα κόστη του προσωπικού και δεν εφαρμόζονται στο ειδικό των ε, του έμεσου κόστους. Περνάμε τώρα στις συστάσεις, ε, που δεν αφορούν μόνο στην Αυστρία, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες. Από τη στιγμή που συντάσσεται ένα σχέδιο ε, κανονισμού, γενικότερου κανονισμού για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ε, είναι ανάγκη να οριστούν επακριβώς και να εξηγηθούν επαρκώς όλες αυτές οι διατάξεις ε, περί απλούστευσης. Η εμπειρία της Αυστρίας υποδεικνύει ότι θα πρέπει να εξετάσουμε σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι διατάξεις αυτές και να τις βελτιώσουμε πριν ε, τις ενσωματώσουμε στον καινούριο κανονισμό που θα υιοθετηθεί για την επόμενη προγραμματική περίοδο ε, σε θέματα πολιτικής ε, συνοχής. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση που αξιοποιούνται διαφορετικά ταμεία, μια προσέγγιση πολλαπλών ταμείων, εάν για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη ε, ε, συνεργεί με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή το ΦΕΟΚΑ, ε, το Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγύσεων, είναι πιο δύσκολο ενδεχομένω να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία η απλουστευμένη. Γίνεται πιο περίπλοκη η κατάσταση και προκαλείται μεγαλύτερη σύγχυση σε όλες αυτές τις διαδικασίες εκαθάρισης. Ε, καλό θα ήταν να έχουμε κατευθυντήριες γραμμές με περισσότερες λεπτομέρειες. Να έχουμε δηλαδή πιο συγκεκριμένες οδηγίες σε τεχνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ενιών. Αυτά όλα τα έχουμε συλλέξει ως προτάσεις από την Αυστρία ε, την προσπάθειά της να ελοποιήσει αυτό το σύστημα. Μπορείτε να ολοκληρώσετε, διακόπτει ο Πρόεδρος. Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε. Μία σύσταση από πλευράς Αυστρίας σε συντομία είναι η εξής. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες εθνικές διατάξεις, για παράδειγμα ισολογισμοί κερδών απολειών, ε, στοιχεία που, οι λογαριασμοί που έχουν ήδη ελεγχθεί από τις τοπικές εθνικές αρχές αν υπήρχε εναρμόνιση των διατάξεων για τις επιδοτήσεις, αυτό θα απλούστευε τη διαχείριση των προγραμμάτων. Ε, έτσι όπως έχει η κατάσταση είναι αρκετά άκαμπτο το σύστημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ. Thank you very much, Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης πολύ για αυτή τη μελέτη που θεωρούμε ότι είναι πολύ επικοδομητική. Είναι μια πολύ καλή ανάλυση των διαφορετικών αυτών ε, θεμάτων που και εμείς παρακολουθήσαμε και για το απλούστευμένο σύστημα όσον αφορά το κόστος. Ωστόσο θεωρούμε ότι ο τίτλος της μελέτης είναι κάπως σύντομος. Θεωρεί μόνο γενικά την απλούστευση. Εμείς σε αυτή τη μελέτη έχουμε την απλούστευση των απλούστευμένων επιλογών κόστους όμως υιοθετήθηκε μια σωστή προσέγγιση επικεντρωνόμενη εσείς σε αυτό το θέμα με ανάλυση σε βάθος. Αληθεύει ότι υπήρξε κάποια κίνηση που είχε κάπως βράδυ χαρακτήρα. Κάποια προγράμματα παίρνουν μεγάλο χρονικό διάστημα για να εγκριθούν. Πρέπει επίση να αναγνωρίσουμε τη διαφορά μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερική Ανάπτυξη. Και εδώ βλέπουμε και το 2009 που χρειαζόταν συγκεκριμένο διάστημα για να ισχύσουν όλα αυτά πάλι και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερική Ανάπτυξη, όπω για το Κοινωνικό Ταμείο. Και βλέπουμε τι ε, διαφορέ που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ένα άλλο σημείο για το Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερική ανάπτυξη είναι ο ετερογενή χαρακτήρα. Έχουμε πολύ περισσότερε μορφέ παρεμβάσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξη που καθιστούν πολύ πιο δύσκολο να καθοριστεί ένα ποσοστό ως ε, flat rate, ως καταποκοπήν ποσό για τις διάφορες δράσει. και Υπάρχει ο πολυσυδής χαρακτήρας αυτών των ε, ε, υπολογισμών ε, στις διάφορες παρεμβάσεις. Είναι ένα περιορισμένο φάσμα όσον αφορά την εμπειρία μας. Εμπειρία πείρα που βασίζεται και στο feedback της προτάσεις, απαντήσεις. Πρέπει να τα δούμε όλα πολύ προσεκτικά και συνετά όλα αυτά ως στοιχεία. Είναι ένα βίωμα που βασίζεται σε κάποιους μήνες όλους και όλους υλοποίησης και για αυτούς τους λίγους μήνες ε, να βασιστούμε σε αυτούς θα είναι δύσκολο σε αυτή τη φάση να πούμε αν θα, είναι, αν θα είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα σε σχέση με αυτό το εύρος ή όχι. Φυσικά προσβλέπουμε στο να υπάρξουν βελτιώσεις και καθότι μπορείτε να δείτε στην πρόταση που υποβάλλεται για το μέλλον υπάρχουν πολλές ε, βελτιώσεις ε, που προβλέπονται. Προσπαθούμε να ενιοποιήσουμε, να εναρμονίσουμε τις εφαρμογές για το απλουστευμένο κόστος μεταξύ των διαφορετικών ταμείων. Επιτρέπουμε την χρήση της δυνατότητας των flat ε, όσον αφορά τις άλλες δράσεις που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα όσον αφορά την ιδιομορφία των ε, ε, πρωτοβουλειών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερική Ανάπτυξης και flat rates όσον αφορά για τα έξοδα στελεχών, για το προσωπικό και τις δαπάνε που συνεπάγονται αυτές οι δράσεις. Ωστόσο, Καταρχήν η βασική προσέγγιση, η ουσιαστική προσέγγιση που υποβάλλεται είναι σωστή και είναι χρήσιμη και για την ανάλυση που πρέπει να γίνει στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα αναλάβω σύντομα την Προεδρία. Εγώ δύο παρεμβάσεις έχουμε. Κύριος Γκάιερ πρώτα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την παρουσίαση που έγινε, για αυτή την μελέτη Το αποτέλεσμα το βρήκα σε σχέση με δύο πτυχές πολύ ενδιαφέρον. Η μία προσέγγιση, η μία σκέψη ήταν αν αυτές οι διευκολύνσεις θα λειτουργούν όπως εμείς το είχαμε φανταστεί και το θέλαμε. Συζητώντας για την επιβάρηση την τελική που συνεπάγεται τον τελικό χρήστη την διοίκηση, ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκολύνσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλει προσπάθειες πραγματικά να διευκολυνθούν και να αλλάξουν αυτές οι κανόνες και κανονισμοί. Το ερώτημα παραμένει, επιτυγχάνεται αυτή η ανακούφιση, η διευκόλυνση που επιθυμούμε. Το αποτέλεσμα είναι μεικτό, είναι ένα μείγμα. Ένα προτέρημα αυτής της μελέτης είναι ότι μας δίνονται επισημάνσεις κάποια στοιχεία σε ποια σημεία υπάρχουν διευκολύνσεις και ότι ίσως δεν επαρκεί απλά κάτι παραπάνω να κάνουμε σε να στρίψουμε μια βίδα λίγο παραπάνω, να κάνουμε δηλαδή μια, να αναλάβουμε μικρή πρωτοβουλία, αλλά χρειάζονται περισσότερες πρωτοβουλίες. Το δεύτερο ερώτημα το οποίο μπορώ να διατυπώσω σε αυτό το σημείο είναι η μεγάλη χρονική καθυστέρηση μεταξύ ενός κανόνα ή κανονισμού που εμείς συντάσσουμε και σύμφωνα με τις απόψεις μας Πιστεύουμε ότι το ίδιο δευτερόλεπτο και όλα θα γίνει πραγματικότητα. Ενώ εντωμεταξύ στην πραγματική εφαρμογή, στην πράξη δηλαδή, στην ευρωπαϊκή καθημερινή πραγματικότητα υπάρχουν καθυστερήσεις. Αυτό και πάλι πρέπει πάντα να το λαμβάνουμε υπόψη ως στοιχείο. Όταν εξετάζουμε την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις των τροποποιημένων κανόνων δημοσιονομικών κανόνων που αλλάζουν και που γίνεται η προσπάθεια να υπάρξουν μεγάλες ε, διευκολύνσεις. Καμιά φορά βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι είναι διευκόλυνση και τι είναι απλουστευμένες διαδικασίες. Αυτό δείχνει ότι μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα πρέπει να ενταχθεί έλεγχος, ελεγκτική δράση, ώστε να δούμε τα, την πείρα που έχουμε συλλέξει, με την πείρα που συλλέξαμε, αν αυτό το οποίο θέλαμε αρχικά επετέφθη ή όχι ο σκοπός. Είναι σημαντική αυτή η επισήμανση, αυτό το στοιχείο. Σε αυτό το σημείο ακριβώς ε, μία ερώτηση θέλω να διατυπώσω μετά από με την ε, ανάγνωση αυτής της μελέτης. Ποιε είναι οι διευκολύνσεις και ποιο επωφελείται από αυτέ. Δεν είναι πάντα το ίδιο πάντα γίνεται, υπάρχει κάποια διαφορά σε αυτό το τελικό χρήστη και όσον αφορά τις, ε, αρχές, ε, τις κρατικές αρχές ή διοικητικές αρχές. Για ποιον κάνουμε εμείς κάποια, θέλουμε να πετύχουμε κάποια διευκόλυνση. Εγώ θα έλεγα για τον τελικό χρήστη. Η διοίκηση είναι η διοίκηση και γραφειοκρατικά και όσον αφορά τις διαργασίες αυτό σημαίνει ότι στην υλοποίηση των προγραμμάτων έχουν ευθύνε οι κρατικές αρχές. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να δυσχεραίνεται και ο βίος τους περισσότερο από την απόλυτα αναγκαίο η επισήμανση όμως ότι η διευκόλυνση αυτή πρέπει να στοχεύει στον τελικό χρήση, χρήστη με που πρέπει να υποφελείται, νομίζω είναι επικοδομητική ώστε να ερμηνευθεί ότι πραγματικά πρέπει να θυμόμαστε ότι για τη διοίκηση, για τις διοικητικές αρχές οποιαδήποτε μεταβολή η τροποποίηση συνεπάγεται επιβάρυνση γιατί ο τυφλοσούρτης που έχουν συνηθίσει αλλάζει και δεν θέλουν οι, ε, οι υπάλληλοι μιας αρχής, μιας διοικητικής αρχής να επιβαρύνονται με τέτοιες αλλαγές ε, τυφλοσούρτη. Η κυρία Γιάλα παρακαλώ. Ο κύριος Γκάιερ είπε αυτά τα οποία ήταν Και ευχαριστώ τους υποβάλλοντες στην εκθέση αυτή, διότι χάρη σε αυτή βλέπουμε ποια είναι τα κυρία σημεία των νέων κανονισμό, κυρίως στον τομέα της ε, νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Άλλα σχόλια από τα μέλη. Εγώ έχω να κάνω ένα σχόλιο. λιγότεροι οργανισμοί, Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. Από τότε που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου εδώ. Πριν από έξι χρόνια η Επιτροπή μας πήρε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει ένα φορέα εκτός Επιτροπής για να μελετήσει το πώς θα έχουμε λιγότερους κανονισμούς. Πρόκειται για μια επιτροπή της οποίας ηγείται ο κύριος Edmund Στόιμπερκ ευθύς εξ αρχής. Την έχετε ακούσει? Μπορείτε να κάνετε κανένα σχόλιο για τη δουλειά που έχει επιτελέσει. Θέλετε... εσείς έχετε κάτι να παρατηρήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα μια ερώτηση να διατυπώσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά που μας αναφέρατε εδώ είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, σίγουρα. Το ερώτημα τίθεται. Πώς συλλήβει συλλογικά αυτά όσον αφορά το κόστος θα καταλήξουν στους νέους κανονισμούς για τα διαδοτικά ταμεία. Με ενδιαφέρει να δω ποιο είναι το τμήμα αυτής της συμφωνία και τι συνεπάγεται. Και πρέπει να το δούμε αυτό, τι επιπτώσεις σε σχέση με τον νέο κανονισμό. Ερώτηση προς την Επιτροπή αυτή. Ευχαριστώ. Uh, Κανείς άλλος δεν το λόγο. Όχι, θα δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα και πάλι στους δύο Σχόλια παρακαλώ. Μελετήσαμε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν μετά από τα πρώτα που κατάληξε η Επιτροπή Στόιμπερ. Κατά την άποψή μας, έγιναν οι πολεμοί και νομίζω ότι τα ωφέλη είναι πολύ μικρότερα από αυτά τα οποία είχαν προβλεφθεί. Και κυρίως αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τα απλοποιημένα ώστε μπορούν να μπορέσουν να μεταφραστούν, αν θέλετε, σε μείωση του κόστου και του διοικητικού. Και είδαμε ότι η μείωση είναι πολύ μικρότερη από αυτή που είχε προβλέψει η μελέτη που έγινε πριν από μερικά χρόνια. Ένα σημαντικό θέμα όμως είναι ότι κάτι το θετικό που μπορεί να γίνει για να πιστούν οι αρχές και τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να κάνουν κάτι συμπληρωματικό στην αρχή για να μειωθεί το διοικητικό. Αυτό είναι να γίνουν ανταλλαγές του τρόπου με τον οποίο εργάζονται οι διοικητικές αρχές. Αν κάποιος δηλαδή είναι πρωτοπόρος σε τέτοιου είδους εμπειρία, θα ήταν εξαιρετικά θετικό εάν μπορούσε να μοιραστεί την εμπειρία. Φερρυπίν, η Ισπανία στην Καστίγια Ραματζά, στην Επιτροπή μας, δεν ξέρουμε πώς δουλεύει το σύστημα. Άρα, προσπαθούμε να δούμε αν κάποιος μπορεί να μας βοηθήσει για το έχω κάνει. Πολύ λίγη βοήθεια όμως παρέχεται το κράτη-μέλη γιατί υπάρχει πολύ λίγη εμπειρία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα ήταν πρακτική σημασία να γίνει κάτι τέτοιο. Βεβαίως οι αρχές έχουν ενδιασμούς για την εισαγωγή του όλου συστήματο, ότι έχουν ακόμη ασάφειε και ερωτηματικά για το πώ ζει το σύστημα. Δεν ξέρω στην Αυστρία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο πώ εμφανίζεται το σύστημα. σω μπορούσαν να υπάρχουν συμπληρωματικά κίνητρα. Διότι νομίζω ότι η αρχή είναι δύσκολη, στο τέλο όλοι θα επωφεληθούμε. Μία φράση μόνο. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσον μπορεί να μεταφερθεί σε άλλους αυτή η εμπειρία. Είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουν ε, με από τους άλλους, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε εάν πραγματικά μπορεί το σύστημα που εισφερώνει σε μία χώρα να το μεταφέρουμε και να το εφαρμόσουμε σε κάποια άλλη. Δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με συνδυασμό κοινοτικής νομοθεσίας και εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή Εγώ είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Επασχόληση, Κοινωνικό Ταμείο. Είδατε η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική. Πριν απαντήσω, θα ήθελα να διορθώσω κανένα δυο σημεία παρουσία. Περίπτωση τη Αυστρία και κυρίω όσον αφορά το Φέντερ. Το Κοινωνικό Ταμείο έχουμε δυνατότητε για τι ε, μη ανοσπληρωμένε από το 2007. Πρόκειται για σύστημα το οποίο εισήγαγε το 2008 το Βέλγιο Φερρυπίν, για να μιλήσει για την πιο Τι μα χώρα εδώ. Τώρα, όσον αφορά το μέλλον. Και ο Ανδρέας θα σας μιλήσει για την παρούσα κατάσταση. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των κρατών μελών σαν αφορά τις αδυναμίες προσπαθήσαμε πρώτα απ' όλα να συνεχίσουμε τα παρόντα συστήματα έτσι ως έχουν, ώστε όσοι είχαν κάνει κάποια επένδυση να μπορέσουν στο μέλλον να επωφεληθούν. Δεύτερον, έγινε πολύ μεγάλη δουλειά όσον αφορά την εναρμόνιση. Έγινε μια παρατήρηση σε σχέση με διαφορετικούς κανόνες μεταξύ των διαφόρων ταμείων. Αυτό είναι μέλος του παρελθόντος, αν εφαρμοστεί ο κανονισμός έτσι ως έχει τώρα. Για ποιο λόγο. Διότι τα τέσσερα ή πέντε ταμεία, ΦΕΝΤΕΡ, κοινωνικό, ε, αλίας, ε, ανάπτυξης υπαίθρου και ε, εγγύσεις έχουν το ίδιο σύστημα και του ίδιου κανόνε βάσει των οποίων θα γίνει η απλοποίηση. Άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με του ίδιου κανόνε το ίδιο σύστημα για τα πέντε αυτά ταμεία. Εκ παραλίλου, η Επιτροπή εισήγαγε επίση την δυνατότητα να γίνει υπολογισμό των διαφόρων συστημάτων που εφαρμόζονται βάσει των παρόντων κανόνων αλλά και βάσει των κανόνων που υπάρχουν από το παρελθόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα το θέμα τη έρευνα Φερρυπίν επιλύεται και αν υπάρχει ανώτατο κατόφλι φεριπίν 40% σε επίπεδο ε, κοινοτικών κανόνων, στο επίπεδο τη έρευνα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το ανώτατο επίπεδο. Και βεβαίω υπάρχει η δυνατότητα να ακολουθηθούν και οι εθνικοί ενισχύοι κανόνε. Εγώ θα ήθελα να πω το εξή για την ε, ανταλλαγές μεταξύ κρατών μελών υπεριφερειών. Η Επιτροπή θέλει να αναπτυχθούν αυτές οι ανταλλαγές εμπειριών μεταξύ κρατών μελών. Και κάναμε με 150 συμμετέχοντες από διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης ε, μία συνάντηση. Έγινε διάλογος μεταξύ των ειδημόνων, διαφόρων περιοχών και της Επιτροπής για την απλοποίηση. Θα ήθελα επίσης να επανέλθω στην ομάδα Στόιμπερ. Στην αρχή της επόμενης εβδομάδας θα υποβάλει έκθεση που αφορά συγκεκριμένα το θέμα αυτό. Θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να επανέλθουμε και να λάβουμε υπόψη την εργασία που επιτέλεσε η Επιτροπή αυτή, προετοιμάζοντας τις προσεχείς νομοθετικές πράξεις μας. Ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω διότι συμμετείχατε σε αυτή την συζήτηση όλους, κυρίως τους εμπειρογνώμονες. Σας ευχαριστώ και τώρα περνάμε στο τελευταίο θέμα που αφορά την ε, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτρικού Συνεδρίου. Παίξαν αποτελεσματικά τα έργα ηλεκτρονική διακυβέρνηση που ανέλαβε στήριξη Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι, διότι είμαι ευρώ σήμερα για να παρουσιάσω την πρώτη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτρικού Συνέδριου στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι, εάν θέλετε, ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ κυβερνήσεων, πολιτών και επιχειρήσεων. Χρειάζεται η χρησιμοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και ε, επικοινωνίας και τεχνικές αλλαγές, αλλά θα πρέπει να γίνει και η κατάλληλη οικονομική έκθεση για να δούμε αν όλα αυτά ε, εφαρμόζονται σωστά. μας, ο οικονομικός μας έλεγχος εστιάστηκε στο περίοδο 2002-2006 για να δούμε κατά πόσον μπορούμε να κάνουμε έλεγχο των επιδόσεων. Τέσσερα κρατημέλη, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Ισπανία επιλέγησαν δεδομένου ότι ο δικός τους ο λογαριασμός ήταν 3 δις του ή 45% των δαπανών του ΕΠΜΑ για τέτοιου είδους προγράμματα κοινωνίας των πληροφοριών. Ε, ζητήθηκε να δούμε εάν τα επιλεγμένα προγράμματα έγιναν σύμφωνα με τις ανάγκες ή αν έπρεπε, αν εφαρμόστηκαν έτσι όπως είχε προβλεφθεί καταρχάς, όπως σε πολλούς άλλους τομείς, τους οποίους αφορούν οι εξελίξεις τεχνολογία, πρέπει να πω ότι βλέπουμε ότι και εδώ οι ανάγκες ε, αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα και από τεχνικής απόψεως και όσον αφορά τις ανάγκες των χρηστών η δυνατότητα χρησιμοποίησης της ηλεκτρονικής κυβέρνησης στα διάφορα κράτη-μέλη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν υπάρχουν οι απαραίτητε δεσμεύσει εκ μέρους των υπευθύνων για να αλλάξουν τα πράγματα. Η περίοδος προγράμματος που ελέγξαμε ε, ήταν αυτή των αρχικών σχεδίων εφαρμογή αυτής της στρατηγική, εκ μέρου των κρατών μελών και είδαμε ότι υπήρχαν κάποια ασφάλματα, αλλά Εάν λάβουμε υπόψη τα συμπράσματα που καταλήξαμε και τα μαθήματα που πρέπει να μάθουμε, μπορούμε να πούμε ότι η πρώτη εφαρμογή του προγράμματο αυτό έγινε με επιτυχία. Είδαμε επίση ότι παρά το γεγονό ότι ε, σχετικά από στρατηγική πλευρά μπορούμε να δώσουμε εύσημα, παρά το γεγονό ότι τα προγράμματα αυτά βελτιώνονται σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν παρόλα αυτά κάποιε αδυναμίε στην στρατηγική, πράγμα που σημαίνει ότι πάντα δεν ε, μπορούσαν να λύσουν τα προβλήματα προτεραιότητα σε αυτά τα προγράμματα. Όσον αφορά τα ίδια αυτά τα προγράμματα, παρά το γεγονός ότι τα παραδοτέα προγράμματα ε, γενικώ παρεδώσαν στις ε, χρονικές περιόδους που είχαν προβληθεί, ε, υπήρχαν πολλές φορές προβλήματα κακού σχεδιασμού ή έλλειψη σωστής μεθοδολογίας εφαρμογής. Ίσως θα πρέπει να δοθούν δυνατότητες ε, καινούριε νέες τεχνολογίες, οι οποίες δεν έτυχαν τις απαραίτητες εκμετάλλευση τότε. Γενικότερα, θετικά, θα μπορούσα να πω ότι τα περισσότερα προγράμματα τα οποία ελέγξαμε από τεχνικής πλευράς ήταν σωστά και οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών ε, για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε δημόσιες ε, ε, δημόσιους οργανισμούς, τους πολίτες και διάφορες επιχειρήσεις γενικά ήταν σωστά. Στην έκθεση κάνουμε κάποιες συστάσεις για να βελτιωθεί ο σχεδιασμός των σχεδίων ε, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο μέλλον, Κάτι το οποίο σημαντικό είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορέσουν να αναπτυχθούν αυτά τα σχέδια διακυβέρνηση, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Γι' αυτό το στόχο, γι' αυτό το λόγο τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν τι κατάλληλε στρατηγικέ που βασίζονται σε στοχευμένε ανάγκε με σαφεί στόχου και να ορίσουν ευθύνε για κάθε ένα από τον εμπλεκόμενο φορέα. Ειδικά στην παρούσα κατάσταση των πραγμάτων, δεδομένου ότι έχουμε λίγους πόρους να διαθέσουμε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η βοήθεια που παρέγεται είναι σωστά στοχευμένη και είναι ε, κάτι το οποίο αξίζει τα χρήματα για τον ε, Ευρωπαίο πολίτη. Τα κράτη-μέλη, θα, έχοντας αυτό υπόψη, θα πρέπει να επιλέξουν τα κατάλληλα προγράμματα και να λάβουν υπόψη την αξιολόγηση που γίνεται. Δεδομένου ότι είναι σημαντικό τα συστήματα που αναπτύσσονται στα διάφορα κράτη-μέλη να μιλούν μεταξύ τους και να συνεργάζονται, το Ελληνικό Συνέδριο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συστάσεις θα επιτρέψουν να υπάρχει διευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα και όλα τα, προγράμματα θα μπορέσουν να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση του ΣΕΤΠΑ. Η ηλεκτρική η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι όλο και περισσότερο επίκαιρη στην καθημερινή ζωή των πολιτών μας. Πιστεύω ότι τα ευρήματα και οι συστάσεις είναι θετικές για τις μελλοντικές εξελίξεις της ε, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και χαίρομαι ότι ο κύριος Μίλντερ στο έγγραφο εργασίας επαναλαμβάνει και χαιρετίζει τις συστάσεις που έχουν γίνει στην έκθεσή μας. Ελπίζουμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικό ε, τρόπο δαπάνης των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων, μείωση του διοικητικού αχθούς και στοχευμένες ενέργεια. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή έχει το λόγο. Chair, uh, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μας για αυτή τη δουλειά η οποία έρχεται στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Οι συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου είναι πάντοτε εξαιρετικά χρήσιμες, πόσο μάλλον εν ώψη της επόμενης προγραμματικής ε, περίοδου το κόστος ανήλθε στα 200 εκατομμύρια ευρώ των δειγμάτων που επέλεξε το ελεγκτικό συνέδριο, που εξέτασε το ελεγκτικό συνέδριο και επέλεξαν τέσσερα κράτη-μέλη. Το δείγμα αυτό έχει να κάνει με έργα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Κάτι το οποίο είναι ένα από τα σκέλη της ε, τεχνολογίας της πληροφορίας και των, ε, της επικοινωνίας γενικότερα βάσει στο ευρύτερο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την ε, Περιφερειακή Ανάπτυξη. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως ε, με τα συμπεράσματα του ελεκτικού συνεδρίου. Τα έργα αυτά δεν έχουν μόνο στόχο την τεχνολογία αυτή καθεαυτή. Θέλουν να ε, κάνουν την υπηρεσία που προσφέρεται πιο επωφελή. Θέλουν να αλλάξουν την οργάνωση ούτω ώστε να υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερα ωφέλη στο μέλλον. Συμφωνούμε με το ελεγκτικό συνέδριο. Ριζικές αλλαγές έχουν σημειωθεί στον ευρύτερο αυτό τομέα τα τελευταία δέκα χρόνια και μάλιστα οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση για την Κοινωνία των Πληροφοριών τελευταία ε, έχουν δραστηριοποιηθεί πολύ προσπαθώντας να συντάξουν ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης ε, για όλα αυτά τα θέματα μέσα στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας. Όλα αυτά είναι ένα εξελίξη. Αυτό που θα ήθελα να πω ε, εν κατακλειδί είναι το εξής. Βεβαίως και θεωρούμε ότι η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Ενισχύεται το μήνυμα που εκπέμπεται και στις προτάσεις κανονισμού που έχουμε υποβάλει εμείς για το μέλλον. Δηλαδή, έμφαση πρέπει να δίνουμε ε, στην επίτευξη των ωφελιών από όλες αυτές τις επενδύσεις. Δεν πρέπει να δίνουμε έμφαση μόνο στην παραγωγή αυτού του συστήματος του τεχνολογικού ε, δεν πρέπει να δίνουμε έμφαση στο τεχνολογικό κομμάτι, αλλά κυρίως στο όφελος που θα αποκομίσουμε από αυτό. Ε, αλλάζουν τα πράγματα πολύ γρήγορα. Πολλά και διαφορετικά μέσα μπορεί η κεντρική διοίκηση να χρησιμοποιήσει, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, για να παράσχει καλύτερες υπηρεσίες. Ε, πολλές προκλήσεις υψώνονται μπροστά μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά και το εξής Το ελεκτικό συνέδριο έχει εξετάσει και το θέμα της αηφορίας και της ε, ε, δυνατότητας διατήρησης ε, του συστήματος σε βάθος χρόνου. Επομένως, το ελεκτικό συνέδριο έχει καταλήξει σε συστάσεις για την διαχείριση του έργου. Θα τις εξετάσουμε εκ του και θα βεβαιωθούμε ότι οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους όλες αυτές τις συστάσεις και θα τις ε, εφαρμόσουν στα μελλοντικά προγράμματα που θα διαχειριστούν. Οι συνάδελφοί μου από την ε, Γενική Διεύθυνση για την Κοινωνία των Πληροφοριών μπορούν να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Ο Πρόεδρος θα έπρεπε να έχουμε ολοκληρώσει τις συνεδρίες στις 11.30. Είναι τώρα 12. Δεν έχουμε χρόνο πολύ. Ε, προτείνω του, στους συναδέλφους σας από την Γενική Διεύθυνση για την Κοινωνία των Πληροφοριών να μας τα υποβάλουν ε, αυτά γραπτός. Θα προσπαθήσω κι εγώ να είμαι σύντομος. Είμαι και εισηγητής άλλωστε για τα θέματα αυτά. Πολύ καλή έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Το ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι όντως η τεχνολογία είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται ραγδαία χρόνο με το χρόνο. θα πρέπει ενδεχομένως να ε, χαρακτεί στρατηγική για κάθε κράτος μέλος, να γίνει σωστή ανάλυση κόστους ωφελιών σε κάθε περίπτωση. Το πιο σημαντικό όμως είναι να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον και να εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές παντού. Πρέπει λοιπόν να διδασκόμαστε ε, ο ένας από τον άλλον, ούτως ώστε όλοι να εξελιχθούμε. Να μάθουμε ε, πράτοντας από αυτά που ήδη έχουν εφαρμοστεί στην πράξη. Δεν θέλω να επεκταθούμε. Κυρία Χέρτσοκ, ωστόσο θέλετε κάτι να πείτε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Σκιώδη, εισηγείται για του σοσιαλιστές να πω και εγώ δύο λόγια. Και η άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή μου, η Ήτρε, είχαμε χθε μόλις μία μήνυα ακρόαση για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και πρέπει εσύ βλέποντας το μέλλον και το παρελθόν να ακολουθήσουμε τη σωστή τροχιά. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη από πλευρά διοίκηση πρέπει να κινηθούν οδηγηθούν προς την 20, στον 21ο αιώνα με αυτές τις τεχνολογίες. Εν τω μεταξύ δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι μόνο 43% των Ευρωπαίων χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως βάση εργασίας. Εδώ και πολύ χρόνο πρέπει για τις, την κάλυψη των αναγκών των Ευρωπαίων πολιτών να μην ξεχνάμε όλες αυτές τις ανάγκες θα πάρουν πολλά χρόνια ακόμα αυτές οι διεργασίες για να καλυφθεί 100% ο αριθμός των Ευρωπαίων. Θέλω να αναφέρω κάποια πράγματα. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ακούγω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν πρόκειται μόνο για τη διαχείριση. Πρόκειται για υπηρεσίες, υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και γι' αυτό θέλουμε να υπάρξει μια μικρή αλλαγή σε σχέση με την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Για μας το output δεν είναι το megabytes και το μέγεθος και η εμβέλεια της τεχνολογίας, αλλά είναι και αυτό συν οι υπηρεσίες που παρέχει η διοίκηση στους πολίτες. Και τα δύο πρέπει να είναι το output ως κύριε δείκτες των επιδόσεών μας και για την ανάλυση κόστους-οφέλους. Θέλουμε επίσης να τονίσουμε ότι πρέπει να κατανοήσουμε την ανάλυση και τις επιπτώσεις σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Να λάβουμε υπόψη και οι ιδιομορφίες των περιφερειών που εμπλέκονται. Υπάρχουν οι περιφέρειες με ιδιαίτερα υψηλή ηλικία των πολιτών τους. Ε, ε, θα είναι διαφορετικό το κόστος λοιπόν από μια περιφέρεια σε σχέση με άλλη τα ωφέλη μπορούν να είναι υψηλότερο το κόστος για να υπάρξουν αυτά τα ωφέλη ανάλογα με τις μειονεξίες ή ιδιομορφίες των περιφερειών. Και σίγουρα πρέπει να συνυπολογίσουμε στην ανάλυση κόστους ωφέλους το κόστος για την κατάθεση επιμόρφωση ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να φτάσουν στο ύψος των περιστάσεων και να χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες όπως πρέπει. Δηλαδή και η κατάρτιση και επιμόρφωση όσων ε, ε, εργάζονται σε αυτό το τομέα και κατάρτιση των πολιτών επίσης ε, για να γνωρίζουν και να έχουν εξοικειωθεί καλύτερα με αυτά. Με τις τροπολογίες αυτές λοιπόν, με αυτές τις παρατηρήσεις για την έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου που έγκαιρα ήρθε σε σχέση με τη συζήτηση της ε, δικτυακής ε, ηλεκτρονικής ημερήσιας διάταξης μπορούμε να προχωρήσουμε. Oh, sorry. Συγγνώμη, μόλις ακούσατε επένους, θέλατε να πείτε κάτι για να ολοκληρώσετε κύριε. Πολύ σύντομα ελπίζω από πλευρά σας. Πολύ σύντομα πρόεδρε, ναι. Σε σχέση με τις προηγούμενες ε, ειδικέ εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, όσον αφορά αρνητικά συμπεράσματα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Στη δική μας έκθεση έχουμε θετική έκβαση γενικά, μια, ένα θετικό τόνο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τα συμπεράσματά μας. Το συμπέρασμα μας λοιπόν είναι σαφέστατο. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τα προγράμματα θα πρέπει να μπορέσουν να προχωρήσουν για την ανάπτυξη των δημοσίων υπηρεσιών στην ηλεκτρονική διάταξη. Κάτι όμως το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτές τις δραστηριότητε, Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλό θα ήταν στην επόμενη περίοδο ως εκκίνηση, ως γραμμή αφετηρία, να μπορέσει να καθορίσει αυτά, να ρυθμίσει αυτά τα στοιχεία τα οποία τονίζουν με αρνητικό τρόπο τα σχόλιά μας στην έκθεσή μας αυτή η ε, έκθεση θα μπορούσε έτσι να συνεισφέρει θετικά για αυτή την επόμενη περίοδο προγραμματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί. Νομίζω επαρκούμε σε αυτά τα σχόλια και είναι θετικό το ότι με αυτόν τον τρόπο για όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη. Είναι η πρώτη έκθεση που είχε θέμα αυτόν τον τομέα θα υπάρξει συνέχεια που θα δοθεί φυσικά, διότι σκοπός μας είναι να δώσουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα στο μέλλον, εν ευθέτω χρόνο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο νομίζω θα μπορέσουμε και περισσότερα συμπεράσματα σε ένα μεγαλύτερο ε, πλαίσιο για όφελος ε, να ε, μπορέσουμε να συναγάγουμε. Σας ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ και είναι το τελευταίο αυτό σημείο στην ημερησία διάταξη για τις σημερινές μας εργασίες. Σας ευχαριστώ όλους. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλή χρόνια σε όλους. Γεια σας. Then we the coordinators meeting. Και τώρα θα ξεκινήσουμε τις συνεδρίες των συντονιστών. Προτού το κάνουμε αυτό, ζητώ όλοι να εγκαταλείψουν την αίθουσα, οι οποίοι δεν ανήκουν σε αυτό το πλαίσιο.